σχέση <clears throat> με την κατάσταση στην Ουγγαρία. Χαιρετίζω την παρουσία του Πρωθυπουργού της ε, Ουγγαρίας, του κ. Βίκτορ Ορμπάν. Καλώς ήλθατε κύριε Όρμπαν. Θα σας πω <clears throat> κύριε και κύριοι πώς θα γίνει η διαδικασία της συζήτησης. Θα δώσω τον λόγο στην Κομισιόν και το Συμβούλιο για να δώσουν τις δηλώσεις τους <clears throat> σε σχέση με το, την κατάσταση στην Ουγγαρία. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους ε, προέδρους ή τους ε, ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων και σε ένα εκπρόσωπο των μη εγγεγραμμένων και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Όρμπαν για να μπορέσει να παρέμβει στα πλαίσια αυτής της συζήτησης και μετά θα συνεχίσει η φυσιολογική διαδικασία συζήτησης. Συμφώνησα με τον κύριο Όρμπαν ότι αν στο τέλος της συζήτησης θέλει να επανέλθει θα πρέπει να μου το αναφέρει και θα του δώσω το λόγο και για μια μονάχα μια φορά στο τέλος αλλά μετά θα έχουν και το δικαίωμα οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων να απαντήσουν στην παρέμβαση του κυρίου Όρμπαν δευτερολογούντες. Και κατά τα άλλα ακολουθεί η διαδικασία ως έχει στο τέλος της, της κανονικής διαδικασίας θα λάβει το χώρο, χώρα και η διαδικασία κάτσει Ερχόμαστε λοιπόν πρώτα στη δήλωση του Συμβουλίου και, και δίνω το λόγο στην κυρία Καλνίνα Λούκασεβίτσκα. Έχετε το λόγο. Uh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τίμερμανς, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ξεκινώ την παρέμβασή μου σήμερα υπενθυμίζοντας τα βασικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο μια οικονομική και πολιτική ένωση που παρέχει στους πολίτες της μια ενιαία αγορά και ελευθερία κυκλοφορίας. Είναι ένωση κοινών θεμελιωδών αξιών. Αυτές οι θεμελιώδεις αξίες καθορίζονται στη συνθήκη και αντικατοπτρίζονται στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και αρχές αυτές περιέχονται επίσης την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ατόμου, στην οποία, την οποία έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άποψη αυτή λοιπόν όλα τα θεσμικά όργανα έχουν τον ρόλο που ορίζουν οι συνθήκες. Το Κοινοβούλιο έχει σημαντικό αξιόλογο ρόλο. Επισημαίνει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή συγκεκριμένες καταστάσεις είναι το βήμα της ευρωπαϊκής πλουραλιστικής δημοκρατίας και για το λόγο αυτό το κοινοβούλιο θεωρούσε πάντα σημαντική τη διαφύλαξη των δημοκρατικών αξιών. Το Συμβούλιο πάντα λάμβανε σοβαρά υπόψη την άποψή σας. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο δεν έχει συζητήσει την κατάσταση στην Ουγγαρία, ούτε έχει συμφωνήσει κάποια θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, θέλω να υπενθυμίσω ότι η Προεδρία και το Συμβούλιο συνολικά προσδίδουν μεγάλη σπουδαιότητα στην ανάγκη διασφάλισης του ότι οι θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης γίνονται πλήρως σεβαστές σε όλη την Ένωση και σε κάθε πολιτική. Η προώθηση της ανεκτικότητας και της διαφορετικότητας είναι η καλύτερη απάντηση στις εξελισσόμενες προκλήσεις ή απειλές για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ε, και τα, τα δικαιώματα του ανθρώπου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, επιτρέψτε μου ταυτόχρονα να, να εκφράσω τι ευχαριστίε μου προ το Κοινοβούλιο, διότι επέτρεψε στι ε, στις Ουγγρικές Αρχές ως άμεσα εμπλοκόμενο ε, μέρος τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Η Προεδρία ευχαριστεί επίσης και τις αρχές της Ουγγαρίας που είναι παρούσες εδώ σήμερα Κύριε Σούλτς, κύριε Τίμερμαντς, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και, κύριε, και, και κύριοι βουλευτές, δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή. Το Συμβούλιο θα παρακολουθήσει προσεκτικά τη συζήτηση και θα προσέξει ιδιαίτερα τις απόψεις που θα εκφραστούν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Καλίνα. Το λόγο έχει τώρα ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν ο κύριος Τίμερμανς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και μέσω εσάς και το Κοινοβούλιο που έβαλε το θέμα αυτό στην μίληση διάταξή του διότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία οδήγησαν σε σημαντικές ανησυχίες. Θα αρχίσω με τη συζήτηση που άρχισε ο Πρωθυπουργό Όρμπαν για την επανεισαγωγή της θανατικής ποινή. Ο πρόεδρος Γιούνκερ και εγώ ήδη κάναμε δηλώσεις επ' αυτού που αποτελούν την επίσημη θέση της Κομισιόν. Το άρθρο της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης απαγορεύει ρητά τι θανατικές εκτελέσεις. Εκτός αυτού, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφασίσει ότι η θανατική ποινή είναι παραβίαση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κατάργησή της είναι προϋπόθεση απαραίτητη για να γίνει κανείς μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δηλαδή είναι τμήμα των κοινών μας αξιών. Για την Κομισιόν τώρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η επαναφορά της θανατικής πηγής θα ήταν αντίθετη με τις βασικές αξίες της Ένωσης. Επομένως θα οδηγούσε στην εφαρμογή του άρθρου 7 της συνθήκης. Οι μηχανισμοί του άρθρου 7 αφορούν τις αξίες που αναφέρει το άρθρο 2 όπως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως γνωρίζετε, οι συνθήκες δεν προβλέπουν την εκδίωξη κάποιου κράτου μέλους. όλα αυτά, το άρθρο 7 προβλέπει ένα μηχανισμό κυρώσεων για να διασφαλιστεί ο σεβασμός και η συμμόρφωση με τις βασικές αξίες που αναφέρει το άρθρο 2. Πιο συγκεκριμένα, για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Θα ήθελα να πω τα εξής. Ο πρόεδρος Γιούνκερ στι 30 Απριλίου δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργό Όρμπαν πρέπει αμέσως να αποσαφηνίσει ότι δεν είναι πρόθεσή του η επαναφορά της θανατική ποινή. Εάν ήταν αυτή η πρόθεσή του, και διαβάζω, τότε θα δημιουργηθεί μεγάλη ταραχή. Η Ουγγρική κυβέρνηση είχε πει ότι δεν, έχει, δεν θα λάβει μέτρα για την επαναφορά της θανατικής πηγής και μας διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός Όρμπαν ότι η Ουγγρική κυβέρνηση θα σεβαστεί όλες τις ευρωπαϊκές συνθήκες στο ακέραιο. Αυτό το είπατε στη συνέντευξη τύπου κύριε Σούλτ στις 30 Απριλίου. Παρ' όλα αυτά, εάν η Ουγγρική κυβέρνηση λάβει μέτρα για την επαναφορά της θανατικής ποινής, θα ήθελα να τονίσω ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει αμέσως όλα τα μέσα που διαθέτει για να διασφαλίσει ότι η Ουγγαρία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος θα συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τον ενωσιακό νόμο και θα σεβαστεί τις ευρωπαϊκές αξίες που αναφέρει το άρθρο 2. Δεν θα διστάσουμε ούτε μια στιγμή. Για τη δημόσια διαβούλευση ως προς τους μετανάστες. Θα ήθελα να κάνω τα εξής σχόλια. Γενικά, η Κομισιόν θεωρεί ότι η δημόσια διαβούλευση μπορεί να είναι σημαντικό εργαλείο διακυβέρνησης για να εφαρμοστούν προγράμματα που έχουν τη στήριξη του λαού. όλα αυτά, επαναλαμβάνω αυτά που είπα και πριν, μια δημόσια διαβούλευση που βασίζεται σε παραπληροφόρηση και σε προκαταλήψεις κατά των μεταναστών δεν μπορεί να θεωρηθεί σωστή βάση για το, τη χάραξη σωστής πολιτικής. Το να συνδεθεί η μετανάστευση με την τρομοκρατία και να θεωρηθούν οι μετανάστες ως απειλή για την απασχόληση των πολιτών είναι απλώς λάθος και θα χειροτερέψει τις προκαταλήψεις. Δεν μπορούμε και δεν θα έπρεπε να κλείσουμε τα μάτια μας στις σοβαρές καμιά φορά προκλήσεις που μας θέτουν τα προβλήματα της μετανάστευσης βέβαια. Αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ τις βασικές μας αξίες και την ανάγκη να διατηρηθεί πλουραλιστική κοινωνία που να βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό και ισοτιμία του καθενός. Η μεταχείριση για όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της πρέπει να αντιμετωπίσουν από κοινού αυτά τα προβλήματα γιατί η Ευρώπη βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό, αλληλεγγύη και ειλικρινή συνεργασία. Χρειαζόμαστε οι πολιτικοί μας ηγέτες να μπορούν να εξηγήσουν στους πολίτες αυτές τις αρχές της Ένωσης δίκαια και ισότιμα και να επιμείνουν στην τήρηση των ευρωπαϊκών αξιών. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προοδεύσουμε στην Ευρώπη, να προχωρήσουμε. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα πράγματα στενά και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συνεχίζει να μας στηρίζει στη σημαντική αυτή προσπάθεια. Ευχαριστώ. Vielen Dank, Herr Ευχαριστώ πολύ κύριε Τίμερμανς για την ομάδα του ΕΛΚ και ο πρόεδρος Βέμπερ. Αξιότιμη κύριε πρόεδρε, κυρία πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρία πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ χαίρομαι για την παρουσία του κυρίου ε, Ορμπάν. Αυτό η παρουσία του δείχνει και το σεβασμό που τρέφει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να τονίσω επίσης ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε ζητήσει να υπάρξει συζήτηση για τη σκανδαλώδη κατάσταση στη Ρουμανία όπου εκατοντάδες χιλιάδες δεν μπόρεσαν να λάβουν ε, μέρος στις εκλογές και η αριστερά πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεώρησε ότι αυτό δεν είναι σημαντικό αλλά παρόλα αυτά έχουμε τον κύριο Όρμαν για πέμπτη φορά εδώ πέρα. Αυτό δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι πάντα έτοιμο να συζητήσει αντίθετα από την αριστερή πτέρυγα αυτού του Κοινοβουλίου. Όταν μιλάμε για την Ουγγαρία, θέλω να υπενθυμίσω ότι η Ουγγαρία είναι και από τις ατμομηχανές της ε, οικονομίας της Ευρώπης με αύξηση 2,8%. που είναι πολύ καλύτερα από πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριστερή κυβέρνηση και ο Βίκτορ Όρμπαν από το 2010 έχει υποστηριχθεί με ένα συντριπτικό σημαντικό ποσοστό 50% και πάλι είναι πολύ πιο μεγάλο ποσοστό αυτό από τα ποσοστά που λαμβάνουν οι αριστερά κόμματα στην Ευρώπη. <clears throat> Έρχομαι τώρα στην Ουγγαρία και το ερώτημα το οποίο τέθηκε. Συζητούμε θέμα, σήμερα το θέμα της στρατικής ποινή. Για μας είναι μια από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές επιτυχίες στην Ήπειρό μας μαζί με άλλα σημαντικά δημοκρατικά δικαιώματα το γεγονός ότι έχει απαγορευτεί η χρήση της θανατικής ποινή και έχει εξοβελιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό τώρα επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό νομίζω ότι είναι απόλυτα βλαβερό για μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει η θανατική ποινή και ζητούμε από τον κύριο Όρμπαν να μην αναλάβει καμία πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή, διότι αυτό θα βλάψει σοβαρά την Ευρώπη. Το δεύτερο θέμα το οποίο τίθεται είναι η αντιμετώπιση της συμμετοχής των πολιτών. <clears throat> είναι σημαντικό ότι ο κύριος Όρμπαν προφανώς εκπροσωπεί τον λαό του, αλλά οι διατυπώσεις που ε, εκφράζει ο κύριος Πρωθυπουργός, αν υπάρχει και στις Βρυξέλλες η ίδια διατύπωση όπως και στη Βουδαπέστη, αυτό έχει ένα εκρηκτικό χαρακτήρα. Είναι πάρα πολλά τα οποία εμεί δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Αλλά, λέω και πάλι στην αριστερή πτέρυγα του Κοινοβουλίου μας, ότι μπορεί να διαφωνούμε για τις εκφράσεις του κυρίου ε, Όρμπαν, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή δύο τρίτα των ετούντων ασύλου στην Ευρώπη δεν ε, εγκρίνεται η παροχή ασύλου και αυτά τα άτομα θα πρέπει να επανέλθουν στις χώρες τους. Σωστά το είπε λοιπόν αυτό ότι πρέπει να γίνει ο κύριος Ορμπάν. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχάσουμε ότι η Ουγγαρία είναι μια χώρα η οποία έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα και η δική μου περιοχή, η ιδιαίτερη περιοχή η έχει να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα στην ε, από πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αιτούνται ασύλου. Όλη αυτή η προβληματική λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολήσει και δεν θα πρέπει να στεκόμαστε στα λόγια αλλά στην ουσία και στην ουσία είναι σημαντικό αυτό το έργο που έχει κάνει και η Ουγγαρία και ο κύριος Ορμπάν. Ευχαριστώ. Για, την, το σοσιαδημοκρατικό Σοσιαλιστικό και Δημοκρατικό Κόμμα, κύριο Πιτέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εθνική διαβούλευση για μετανάστευση και τρομοκρατία ως αν τα δύο φαινόμενα ήταν συνδεμένα. Η επίκληση της θανατικής ποινής ε, ως ε, προληπτικό μέτρο, ως ε, η πρόκληση σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μιας πιθανής ανελεύθερης δημοκρατίας όπως σωστά ανέφερε ο κύριος Τίμεμαντς είναι μόνο κάποια από τα πρόσφατα κείμενα και θέσεις του κυρίου Όρμπαν. Η συζήτηση πρέπει να είναι σαφής δεν προκύπτει από προκατάληψη κατά του κυρίου Όρμπαν ή από αντιπάθεια για το γεγονός ότι ο κύριος Όρμπαν ανήκει σε άλλη πολιτική οικογένεια από αυτήν στην οποία ανήκω εγώ. από μια προσπάθεια να, να, κάνουμε μαθήματα. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Όρμπαν με την δηλώσει του αυτές ξεπέρασε τα όρια της αξιοπρέπειας. Κάτι που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Είπε ο κύριος Βέμπερ ότι τα προβλήματα δεν λύνονται φορτώνοντας τα προβλήματα σε άλλους που έχουν διαφορετικό πολιτικό ένδυμα. Εγώ επαναλαμβάνω, το δεν τίθεται το θέμα επειδή ο κύριος Όρμπαν ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το οποίο σέβομαι απόλυτα, αλλά διότι βλάπτει τις βασικές αξίες πάνω στις οποίες είναι θεμελιωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το, σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει έκπτωση. Η Ουγγαρία, στην Ουγγαρία το πρόβλημα δεν είναι επίθεση στη δημοκρατία με το κλασικό τρόπο που γνωρίζουμε, αλλά η ε, το άδειασμα της δημοκρατίας όπως το γνωρίζουμε το οποίο μπορούμε να το πούμε με πολλούς τρόπους ε, λέξεις, δημοκρατία, ελευθερία γίνονται κενά σλόγγαν και χωρίς, και χωρίς περιεχόμενο γίνεται ένα κράτος σύγχυσης ένα, όπου η δημοκρατία γίνεται ένα θέαμα χαμηλού επίπεδου ένα παιχνίδι λασπολογίας επαναφέροντας τις ακραίες δυνάμεις κάτι που πρέπει να ανησυχεί όλους μας ναζιστικές φασιστικές δυνάμεις. Αυτό ανησυχεί ιδίως, όχι η βαρύτητα των δηλώσεων, αλλά το σκοτεινό αποτέλεσμα που δημιουργούν αυτές οι δηλώσεις. Φτάνουν αυτή τη στιγμή οι απειλές θανάτωσης ενός ε, ε, ομοφιλόφιλου ακτιβιστή στη Βουδαπέστη που θέλω να, για τον οποίο θέλω να εκφράσω την πληρελεγγύη μου από τις προκλήσεις, οι προκλήσεις αυτές ωστόσο πιστεύω ότι είναι όπλα παραπλάνησης της μάζας ε, προσπαθεί να αποστρέψει την προσοχή των Ούγγρων πολιτών από τα πραγματικά προβλήματα που ζει η Ουγγαρία οικονομικά και κοινωνικά σοβαρότερα προβλήματα κλείνω εγώ κατανοώ και αγαπώ τον Ουγγρικό λαό ως ε, Ιταλός θυμάμαι όταν την εποχή που ο δικός μας Πρωθυπουργός υπονόμευε την αξιοπιστία και της χώρας μας. Πιστεύω κύριε Όρμπαν ότι δεν πρέπει να κάνετε το ίδιο εσείς. Η Ουγγαρία είναι μια μεγάλη χώρα, αξίζει καλύτερο. Δεν μπορεί να γίνει ένα παλκοσέλνικο όπου επιτρέπονται τα πάντα και όπου οι αξίες της κοινή συνύπαρξής μας γίνονται κομμάτι ενός παιχνιδιού για να πάρετε κάποιες ψήφους. Και αν δεν έχετε σεβασμό προς τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχετε ε, σεβασμό στην αξιοπρέπεια του λαού σας. Meine Damen und Herren, ich um <coughs> Σας ζητώ συγγνώμη. Υπάρχει ένας συνάδελφος ο οποίος θέλει να σας θέσει, ήθελε να σας θέσει ένα ερώτημα. Εγώ δεν πρόλαβα και έδωσα το λόγο στον κύριο Πιτέλα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να αποδεχτείτε αυτή την ερώτηση. Κύριο Σουελίνη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βέμπερ, εγώ σας σέβομαι και το πρόσωπό σας και τα λόγια σας. Είσαστε ο πρόεδρος της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σας ρωτήσω ότι πιστεύετε για την εξή πρόταση. Η Ευρώπη δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα διαλυμένο σύστημα θεσμών που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν κάνουν αυτό το οποίο δημιουργήθηκαν να κάνουν δεν είναι πια μια κοινότητα αξιών. Όχι, αυτό δεν το λένε οι εξτρεμιστές. Αυτή είναι παράθεση από ένα από τους ηγέτες του Φίντες πρόσφατα, κύριε Βέμπερ. Συμφωνείτε με μια τέτοια αντιμετώπιση. Θεωρείτε ότι δουλεύετε σε ένα διαλυμένο όργανο. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες απόψεις δυστυχώς στην Ευρώπη ακόμα και στη σοσιαλιστική ομάδα και σε άλλες πολιτικές οικογένειες υπάρχουν άτομα τα οποία εκφράζουν τέτοιες απόψεις. Αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα είναι πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα με τις Ουγγαρίας και σας λέω ότι είναι μία από τις πρωτοπόρες χώρες της Ευρώπης σε οικονομικό επίπεδο και ότι οι πολίτες της Ουγγαρίας είναι προφανώς ικανοποιημένοι με τους ηγέτες τους και τους έχουν υποστηρίξει σε δημοκρατικές εκλογές. Εντάξει, για να απόλυτη ισότητα. Η κυρία Γκάλ Πέλση ήθελε να θέσει σε εσάς κύριε Πιτέλα μια ερώτηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν δέχεστε αυτό το ερώτημα. Κυρία Γκάλ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Πιτέλα, αλλά επειδή έχω το λόγο θα το κάνω αυτό για να υπάρξει ισορροπία. Κύριε Πιτέλα, μια στιγμή λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη, κύριος Γκάλερ ήθελε να λάβει το λόγο και όχι η κυρία Γκάλ Πέλς. Στη συνέχεια μπορείτε να λάβετε το λόγο, λέει, στην κυρία Γκάλ Πέλς, ο πρόεδρος. Παρακαλώ. Όχι, κυρία Γκάλ μπορείτε να συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσω λοιπόν τότε. Τα πράγματα γίνουν λίγο πιο περίπλοκα. Κύριε Πιτέλα, τι άποψη έχετε ο κύριος Τίμεμανς μας απείλησε στην πράξη. Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει το άρθρο 2. Δεν είστε υπέρ της ανοιχτή συζήτηση των προβλημάτων κύριε Επιτέλα, υπάρχουν θέματα ταμπού. Αν έχετε κάποιο τέτοιο κατάλογο να μας τον δώσετε, γιατί αλλιώς δεν ξέρω σε τι κοινοβούλιο βρίσκομαι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη θανατική ποινή. Είναι ταμπού αυτό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα προβλήματα της μετανάστευσης. Ταμπού είναι και αυτό. Τι μπορούμε να συζητήσουμε. Ποια, πού είναι ο κατάλογος των απαγορευμένων θεμάτων. Συνάδελφε να σας πω τι, τι άποψη έχω για τον κύριο Τίμερμαν. Έχει, τον εκτιμώ απόλυτα, τον θεωρώ φίλο και τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και εκτιμάται πολύ περισσότερο από μένα μόνο και το Κοινοβούλιο. Δεν ε, απλοποιούμε τη συζήτηση. Προφανώς μπορούμε να συζητήσουμε τη μετανάστευση. Το κάνουμε και εμείς συνεχώς έχουμε διαφορετικές απόψεις. Το πρόβλημα είναι ότι τίθεται σε, τίθενται σε συζήτηση βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη εφαρμογή της θανατικής ποινής είναι μια θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ένας επικεφαλή κυβερνήσεω, που δεν είναι ένα απλό πολίτης που βρίσκεται ε, σε ένα καφενείο και κουβεντιάζει λέει ότι θέλει να καταργήσει την κατάργηση της, ε, να επαναφέρει τη θανατική ποινή σε μια χώρα είναι ένα θέμα που πρέπει να μας ανησυχήσει. Δεν είναι κάτι ασήμαντο. Ο αρχηγός μιας κυβέρνηση, ε, μιας χώρα της Ένωση, όταν μιλά για μια ανελεύθερη δημοκρατία δεν πρέπει να μα ανησυχήσει. Δεν το λέει κάποιο ε, σε ένα καφενείο. Ο επικεφαλή μία από τι 28 κυβερνήσει τη Ένωση το λέει. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. Κάτι πρέπει να το κάνω σαφέ. Όταν ο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι υπάρχει μια παραβίαση του άρθρου 2 και πρέπει η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει το άρθρο 2, αυτό δεν είναι μια απειλή, είναι μια διαπίστωση πραγματικότητας. Και δεν μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε αυτό που είπε η κυρία Γκάλ Ο κύριος Κίρκοφ έχει το λόγο τώρα για δύο λεπτά για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Uh, uh, Πρόεδρε και Αντιπρόεδρε κύριε Υπουργέ. Ως μέλη της Ένωσης συνυπογράψαμε μία σειρά βασικών αξιών και αρχών για τους πολίτες. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις, αλλά εμείς στο Κοινοβούλιο είμαστε ένα βήμα συζήτησης και πολλές φορές και πρότασης λύσεων. Αν όμως θέλουμε να γίνουμε δίμιος και δικαστής για όσους διαφωνούν, τα πράγματα αλλάζουν. Εδώ μιλήσαμε για προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για την εφαρμογή των συνθήκων. Αλλά το γεγονός είναι ότι η αριστερά του Κοινοβουλίου εδώ επιτίθεται ακόμη μια φορά στην κεντροδεξιά γιατί μερικές χώρες μέλη τολμούν να μιλήσουν για θέματα που ενδιαφέρουν τους εκλογεί του. Υπάρχει το δικαίωμα να συζητιούνται τέτοια πράγματα ακόμη και αν δεν είναι από τον κατάλογο των προεγκεκριμένων θεμάτων κύριε Πιτέλα. Γιατί πρέπει πάντοτε να θεωρούμε ότι το βήμα είναι μεταξύ Κοινοβουλίου και κάποιου κράτους μέλους αντίθεση. Εδώ στην Ένωση υποτίθεται ότι είμαστε όλοι εταίροι, όχι δικαστές σημαίνει τον δε. Ο λαός της Ουγγαρίας και οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν θέλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα να γίνουν πεδίο μάχης κομματικών αντιπαραθέσεων. Γίνονται συζητήσεις μεταξύ Κομισιόν και Ουγγρικής Κυβέρνησης όπως είναι και το σωστό. Συζήτηση έχει γίνει στην Επιτροπή Εσωτερικών Πολύ σωστά και αυτό. Αλλά αναρωτιέμαι, γιατί είμαστε σήμερα εδώ, γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή δεν θα οδηγήσει πουθενά. Δεν θα ωφελήσει κανέναν μάλλον. Κύριε Κύρκοπ, υπάρχει χαλάζια κάρτα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κίρκοπ, θα θέλατε ο Πρωθυπουργό της χώρας σας να δηλώσει ότι θέλει να οικοδομήσει ανελεύθερη δημοκρατία. Θα συμφωνούσατε με τον Πρωθυπουργό σας αν έλεγε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα, αλλά των εκλογέων. Και παρομοίως είναι θέμα τέτοιο και να μιλήσει ο λαός της Ουγγαρίας, η εκλογής του ηγέτη που εξέλεξαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους και δημοκράτες, η κυρία Ιντφέλτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η παρουσία του Πρωθυπουργού κύριου Όρμπαν εν γέννη είναι ευπρόσδεκτη στο Κοινοβούλιο. Ελπίζω όμως να μην τον απογοητεύσω αν δεν ασχοληθώ πολύ ε, μαζί του, διότι η συζήτηση δεν αφορά τον ίδιο. Η μη δήλωση του Συμβουλίου δείχνει την ηθική χρεοκοπία του Συμβουλίου και το γεγονός ότι είσαστε τελείως μακριά από τις συνθήκες. Ναι, συνάδελφοι, μπορεί να κάνουμε μία συζήτηση για τη θανατική ποινή και μπορεί να είναι πολύ σύντομη. Εγώ την απορρίπτω απόλυτα, η ομάδα μου την απορρίπτει, δεν έχει θέση στην Ευρώπη, δεν έχει θέση στην Αίγυπτο, δεν έχει θέση οπουδήποτε στον κόσμο. Τέλος συζήτησης. Ωστόσο, το θέμα της θανατικής ποινή είναι μια προσπάθεια να απομακρυνθούμε από το πραγματικό και πολύ πιο σημαντικό θέμα, τη, με, την πολιτική μετανάστευση. Και αυτό δεν είναι μια γνώμη, είναι πολιτική τη κυβέρνηση. Τι κάνει λοιπόν η Επιτροπή, Ξεκίνησε μια νομική ανάλυση τη συμβατότητα τη νέα νομοθεσία με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συμφωνεί με τι με τις ε, πολιτικές μετανάστευση και σύλλου της Ένωσης. Η Επιτροπή έχει ευθύνη να δράσει. Συμφωνώ με την κριτική προσέγγιση σας, θα περίμενα ωστόσο περισσότερα από την Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Άκουσα τον κύριο Βέμπερ. Είναι σαφέστατο σε μένα ότι το ΕΡΚ μπορεί να χρησιμοποιήσει επικριτικές φράσεις, αλλά είστε ακριβώς υποστηρίζετε απόλυτα τον κύριο Όρμπαν και τις θέσεις του. Είναι σαφές λοιπόν πού βρίσκεται τώρα ε, ε, το ΕΛΚ. Δεν απορρίπτει, δεν τις θέσεις του κύριου Όρμπαν. Η κατάσταση στην Ουγγαρία δείχνει την ανάγκη να έχουμε γρήγορα ένα μηχανισμό παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη στήριξη του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ εδώ μαζί σας κύριε Βέμπερ. Πρέπει να καλύψουμε το κενό μεταξύ του άρθρου 7 που είναι η πυρηνική λύση Αφενό και άλλων μορφών νομική δράση αφετέρου. Γι' αυτό εμεί υποστηρίζουμε ένα δημοκρατικό σύμφωνο. Ξέρω ότι και άλλοι εξορτάζουν μηχανισμού για την εφαρμογή των θεμελιώδων δικαιωμάτων. Το χρειαζόμαστε. Ξέρω κύριε Τίμερμαν ότι είπατε πω τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν ποσοτικοποιούνται, δεν μετρούνται με δόσεις. Μπορούν όμως πιστεύω και το Κοινοβούλιο ως κοινό εγχείρημα θα έπρεπε να ετοιμάσει προτάσει για έναν τέτοιο μηχανισμό. Ελπίζω ότι θα είναι μαζί μας η Επιτροπή για να προωθούμε τις θέσεις που θεωρούμε όλοι σημαντικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ιντ Φέλντ. Ο κύριος Σέλεριτς θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα. Δεν σας εκπλήττει αυτό. Κύριε Έλεριτς, συμφωνείτε, έχετε το λόγο. Είναι η πρώτη ερώτηση που θέτω αυτή τη βδομάδα. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Μου με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συνολική σας απόρριψη της θανατικής ποινή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει αυτό ότι δεν πιστεύετε σε μια πλήρη δημοκρατία. Τι γίνεται αν ένα κοινοβούλιο εκφράσει την ε, θέληση του λαού και πει ότι θέλει να υπάρξει στρατηγική ποινή. Πιστεύετε ότι και πάλι δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα είναι πολύ σαφέ, λέει η κυρία Ινφελτ. Αν οποιαδήποτε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαναφέρει τη θανατική ποινή, έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν για κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορούν συγχρόνω να είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα αυτό είναι απόλυτα σαφέ. Ευχαριστώ. Για την ε, Ενωμένη ΕΕ, Ευρωπαϊκή Αριστερά, η κυρία Βεργιά, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μια ακόμα φορά συζητούμε την κατάσταση στην Ουγγαρία. Ακούμε τις ίδιες φωνές στο ημικύκλιο. Σίγουρα ο κύριος Σορμπάν θα μας πει ότι και άλλοι έχουν μια αντιμετώπιση παρόμοια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό, και αυτό δεν εξαρτάται από το πολιτικό του χρώμα. Παντού παίζουν με το λαϊκισμό κυβερνήσεις στην ε, Ουγγαρία έχει συμπυκνωθεί ο κατάλογος όλων αυτών των πραγμάτων που δεν πρέπει να κάνει κάποια χώρα. Μετά από τον Οκτώβριο και τη συζήτηση την προηγούμενη, τόνισε η Amnesty International ότι είναι χωρίς προηγούμενο οι καταδιώξεις των ΜΚΟ. Υπάρχει ένας πολιτικός λόγος που στέλνεται κατά των Εβραίων, κατά των ομοφιλοφίλων, κατά των ετούν, των ασύλου κτλ. Υπάρχει αυτό το ερωτηματολόγιο το οποίο συνδέει την μετανάστευση με την τρομοκρατία. Υπάρχουν οι δηλώσει για θανατική πονή. Όπως ε, <clears throat> ζητήσαμε λοιπόν και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να γίνει αυτή η συζήτηση. Αυτό έγινε γιατί ο κ. Σόρμπαν είπε ότι θα πρέπει το θέμα τη θανατική ποινή να γίνει εθνική αρμοδιότητα. Και αν δεν λειτουργούσε η προστασία των πολιτών χωρί θανατική ποινή, θα πρέπει να επαναφερθεί η θανατική ποινή. Μέχρι πού θα φτάσουμε χωρί να αντιδράσουμε σε όλα αυτά. Το άρθρο 7 είναι ουσιαστικά μία φενάκι. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αποτροπής. Μία διαδικασία επιπαραβάση, ακόμα και αυτή, είναι αμφίβολη αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δράσουμε και εναντί της Ουγγαρίας αυτή τη στιγμή. Αλλιώς τι νόημα έχει το άρθρο των συνδικών μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φερισιά. Για τους πράσινους έχει η πρόεδρος Ρεμπέκα Χάμς. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι σχεδόν όλα έχουν λεχθεί και έχει τονιστεί η φρίκη που νιώθει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Ορμπάν και αυτά που ελέγχθηκαν για τη θανατική ποινή. Είναι αλήθεια ότι σήμερα το 2015 κάποια ευρωπαϊκή κυβέρνηση θέλει να επαναφέρει τη θανατική ποινή. Θα ήταν έτοιμη να το κάνει. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θα ήθελα να σας θέσω κύριε ε, Όρμπαν γιατί πολλοί από εμά θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι και το τέλος μιας παρουσίας μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο θέμα είναι το ερωτηματολόγιο για την πολιτική της, ε, για τη μεταναστευτική πολιτική και το ύφος, η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτό το εραυματολόγιο. Αυτό σίγουρα δεν συμβάλλει στο να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα τη μετανάστευση που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και των προσφύγων πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ουσιαστικά αναμόχλευση παθών και παρακίνηση σε μίσο. Η, η Γερμανία είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την έννοια τη, του δηλητηριασμού των απόψεων. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε μονάχα για τον Βίκτορ Όρμπαν και την Ουγγαρία. Μιλάμε για μας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή όταν ένα κράτος μέλος θέλει να αποστραφεί από τις βασικές αξίες και αρχές που απεδέχθη όταν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται όταν ένα κράτος μέλος δεν θέλει να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία έχουμε συμφωνήσει όλοι για μένα. Δεν μπορεί να προχωρήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα κάτω από τέτοιες συνθήκες όταν δεχόμαστε να παραβιάζονται αυτά τα δικαιώματα και όλα αυτά θυσιάζονται στον ε, βωμό μιας πολιτικής συμφερόντων. Αλλιώς θα έχουμε τα εθνικιστικά ρεύματα τα οποία θα οδηγήσουν στην καταστροφή τους. Καταστροφή της στο ευρωπαϊκό όραμα. Κατά τη δική μου άποψη είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην γονατίσει όπως έκανε η Λεπτονική Προεδρία, είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό όχι μόνο στην Ουγγαρία, αλλά και με άλλα κράτη-μέλη, οποιαδήποτε προβλήματα τα οποία τίθενται για την ελευθερία του τύπου, παραδείγματο χάρη, όπως κάναμε και στο παρελθόν, να τονίσουμε τους μηχανισμούς που είναι απαραίτητοι, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε μοναχά τα θέματα της οικονομικής σταθερότητας και του προϋπολογισμού, αλλά να μπορούμε να διατηρήσουμε στην Ευρώπη την προάσπιση των αρχών που έχουμε θεμελιώσει και που σήμερα και το τέλος της βαρβαρότητας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, να μπορέσουμε επιτέλους να εγγυηθούμε για αυτές τις αρχές στους πολίτες μας. Είδαμε ε, την καταπίεση από τις αστυνομικές δυνάμεις στην Ισπανία. Νόμιζα ότι ήταν ένα αστυνομικό κράτος. Τελείωσε ο χρόνος σας, λέει ο πρόεδρος. Όλα αυτά τα οποία βλέπω με έχουν κλονίσει ιδιαίτερα. Θα πρέπει να αλλάξω αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Θα πρέπει να τηρηθούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα πλήρως στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Κατσοντεμπέσκι θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα, κυρία Χάπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι προς την κυρία Άρμς και έχει ως εξής. Μιλήσατε με πολύ ωραίο τρόπο για αξίες, για την διαβούλευση για τους μετανάστες. Γιατί δεν γίνεται συζήτηση τόσο συγκινησιακή για το τι γίνεται στη Γερμανία. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε ότι υπάρχουν σπίτια που καίγονται, διαδηλώσεις ε, μεταξύ του πληθυσμού σε πολλές πόλεις. Ξέρετε την κατάσταση στη Γερμανία. Ξέρετε τι γίνεται στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή δεν δέχονται τους μετανάστες. Και αυτό θα πρέπει να αποτέλεσμα αντικείμενο μια συζήτηση. Δεν βλέπω όμω κανένα να θέλει να συζητήσει. Δεν γίνεται συζήτηση για το τι γίνεται στη Γαλλία ή τη Γερμανία. Αντίθετα, άλλο η Ουγγαρία. αν παρακολουθήσετε τη συζήτηση στη Γερμανία, θα δείτε ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχουν λάβει χώρα στην Γερμανία θα διωχθούν βάσει του δικαίου και της δικαιοσύνης. Η Γερμανία κρατάει μια ανοιχτή πολιτική για τους πρόσφυγες και υποστηρίζει την αρχή των ποσοστώσεων κατόπιν εορτής πιστεύω εγώ αλλά εν πάση περιπτώσει την υποστηρίζει. Ακόμα και σε ό,τι αφορά την πολιτική προσφύγων η Ευρώπη. Κυρία Χάρμς, δεν πρέπει να, συνεχί... δεν πρέπει να ξεπερνάτε το όριό σας. Απαντήστε στο ερώτημα για την ομάδα των, ε, της e κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το να βάλουμε στη μέση διάταξη την θανατική ποινή να πούμε ότι οι ανελεύθερε δημοκρατίε είναι επιτυχία και λειτουργούν καλύτερα από τι δημοκρατίε και πρέπει να είναι μοντέλα προ υπόδειγμα. αυτέ είναι οι τελευταίε δηλώσει του Πρόεδρου Όρμπαν που δεν αφήνουν χώρο στη φαντασία και προστίθενται σε νόμου που φημώνουν την ελευθεροτυπία, που υπονομεύουν την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών και που στερούν τον εγγυητικό ρόλο του συνταγματικού δικαστηρίου. Επιπλέον ξεκίνησε, σαν να μην αισθανετά όλα αυτά, μία μεροληπτική ε, διαβούλευση για τα θέματα της μετανάστευσης. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι το DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό εξασφαλίζεται για τα κράτη-μέλη όχι μόνο τη στιγμή της προσχώρησης αλλά και εκ των υστέρων. Είναι απαράδεκτο να αποδεχόμαστε αυτή την παρέκβαση κατά της Δημοκρατία στην Ευρώπη και να ε, βάζουμε το κεφάλι μας στην άμμο όπως η Θοκάμιλι. Όλοι πρέπει να δράσουν από την Κομισιόν και μετά που πρέπει να προχωρήσει στην παρακολούθηση ε, του σεβασμού των δικαιωμάτων ανθρώπου χώρα προς χώρα. Όσοι εισηγήτρια για τα το σεβασμό των θεμελιών δικαιωμάτων στην Ένωση έχω προτείνει έναν πιο εξελιγμένο μηχανισμό παρακολούθησης της, του σεβασμού με δράσεις ε, που θα πρέπει να αναλαμβάνονται για την πλήρη υλοποίηση των αρχών ε, και δικαιωμάτων που εξασφαλίζει ο χάρτης. Πρέπει να υπάρξει και μια τράπεζα δεδομένων για την κατάσταση των θεμελιών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη, σε κάθε κράτος μέλος και να διευρύνουμε το πλαίσιο αξιολόγησης του Δικαστηρίου της Ένωσης και στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων από κάθε και του κράτους δικαίου από κάθε κράτος. Όλα αυτά για να αποφύγουμε να γίνει ο κίνδυνος πραγματική παραβίαση όπου συμβαίνει ή θα συμβεί σύντομα στην Ουγγαρία. Σήμερα δεν μιλάμε για δηλώσεις ενός αφελούς πολιτικού που χρησιμοποιεί δηλώσει ω προπαγάν, εργαλείο προπαγάνδα, αλλά ενό πρωθυπουργού που δεν είχε κανένα πρόβλημα να αλλάξει το σύνταγμα τη χώρα του για να το κάνει να σεβαστεί την λαϊκιστική και ανελεύθερη προσέγγιση που θέλει να ακολουθήσει. Είναι πολύ, πρέπει να δράσουμε τώρα πριν, πριν είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ κύριε Φεράριο. Ο κύριο Ζάιρ θέλω να σα θέσει ένα ερώτημα. Το αποδέχεστε, παρακαλώ κύριε Ζάιρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα πάρα πολύ σύντομο ερώτημα. Γιατί σας σοκάρει να υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση για ένα σημαντικό θέμα όπως είναι η πολιτική μετανάστευση όταν θέλουμε να ξέρουμε την άποψη όλων των ε, πολιτών της Ουγγαρίας. Αυτό που μας σοκάρει δεν είναι ότι γίνεται μια διαβούλευση, αλλά το αντικείμενο της διαβούλευσης. Από τη στιγμή που ένα κράτος μέλος, ο Πρωθυπουργός ενός κράτου μέλους, ξεκινά μια δημόσια διαβούλευση για την επανεισαγωγή της θανατικής ποινή, σημαίνει ότι γυρίζουμε στο οφθαλμό αντιοφθαλμού, στις πρωτα, πρωτόγονες ε, νομοθεσίες. Αυτό είναι που σοκάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία είναι βάση της ε, ύπαρξης της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για τους μη εγγεγρα... έχει εγγεγραμμένους Μπαλτσό. Όταν είδα στην ημερήσια διάταξη ότι θα μιλούσαμε για την κατάσταση στην Ουγγαρία, δεν κατάλαβα γιατί. Ως εκπρόσωπος του Γιόμπικ δεν είχα ακούσει ότι έγινε τίποτα στην Ουγγαρία που να δικαιολογούσε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Τώρα μας μου δείξατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν σέβεται τις αρχές που διακηρύσει, τις αρχές της ελεύθερης έκφρασης ας πούμε. <clears throat> Γιατί να μην γίνει δημόσια συζήτηση για τη μετανάστευση σε μια χώρα μέλος. Γιατί να μην μπορούμε να θίξουμε τα ταμπού αν θέλει να το κάνει η κοινωνία. Θέλετε να μας ε, προκαθορίζετε ποια θέματα, με ποια θέματα θα ασχολείται κάθε κυβέρνηση και τι θα λέει στους πολίτες αν η κυβέρνηση Ουρμπάν ακολουθήσει την οδό που άρχισε η Ουγγαρία μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας τότε δεν υπάρχει πρόβλημα οδηγούμεθα προς Ομοσπονδία και το Φίντες ακολουθεί αυτό την οδό ως μέλος του ΕΛΚ ο πρόεδρος Μπαρόσο δήλωσε στον κύριο Όρμπαν μετά την ε, Ουγγρική Προεδρία ότι η Ουγγαρία τα πήγε καλά και κατάφερε σημαντικά πράγματα. Επομένως, αφού δηλώθηκε ότι είναι τόσο σημαντική για μας και η ακαιρεότητα της Ουγγαρίας, καταλαβαίνετε ότι στην Ουγγαρία δεν γίνονται μόνο αρνητικά πράγματα. Υπάρχει μια ερώτηση της κυρίας Ιώτη προς εμάς. Συμφωνείτε να απαντήσετε, κύριε Ιώτη. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένας πρώην βουλευτής, Γιώργη Γιούλα Γιαζίβα γίνεται, του κόμματός σας, που απείλησε μία, μία νέα γιατί είναι ακτιβιστής ε, γκέι η οποία ζει από τον περσμένο Ιούλιο υπό την απειλή τη ζωής της. Υπάρχουν ε, κάποιοι που προσφέρουν 10.000 ευρώ για το κεφάλι της. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό, Θέλετε, θα, θα καταδικάσετε αυτή την πρώην συναδελφό σα. Θα ήθελα να ξέρω τι, ποια είναι η άποψή σα. Κύριε Μπάλτσο. Ίσως. Το Ιόμπικ Μπορείτε να πείτε το Ιόμπικ έχει στραφεί εναντίον των ομοφιλοφίλων στην Ουγγαρία, αλλά δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έχω δει καθόλου ειδήσει προ την κατεύθυνση αυτή. Δεν ξέρω από πού βρήκατε αυτήν την ιδέα, δεν ξέρω από πού δημιουργήσατε αυτή την εικόνα. Το Γιόμπικ δεν έχει ποτέ απειλήσει κανένα με τέτοιο τρόπο στην Ουγγαρία. Αυτό το οποίο μπορεί να είπαμε ήταν ότι η προπαγάνδα υπέρ της ομοφιλίας δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να συμβεί στην Ουγγαρία. Δεν πειράξαμε όμως και δεν απειλήσαμε ποτέ κανένα εκεί. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Πρωθυπουργό του κ. Όρμπαν, αλλά προηγουμένως μία διευκρίνηση. Στον πρώτο αυτό γύρο υπήρξαν πολλές ερωτήσεις που ε, να γίνουν. Φυσικά δεν θα έχουμε το ίδιο την ίδια διαδικασία στο δεύτερο γύρο γιατί θα ξεφύγουμε τελείως από το χρόνο μας. Δίνω λοιπόν το λόγο στον Πρωθυπουργό κύριο Ορμπάν. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, ήλθα εδώ διότι συζητάτε την κατάσταση της χώρας μου, της Ουγγαρίας. Είναι πάντα μία τιμή και μία χαρά να δω ότι ενδιαφέρεστε για θέματα που έχουν να κάνουν με την Ουγγαρία. Όταν λοιπόν τίθεται το θέμα της Ουγγαρίας, εγώ είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω εξ ονόματος της χώρας μου και του λαού μου. Οι Ούγγροι αποφάσισαν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα δημοψήφισμα. Είμαστε ακόμα υπερήφανοι για την απόφαση αυτή να γίνουμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί είναι λογικό να έχω έρθει εδώ γιατί η Ευρώπη θέλει να δει και πώς έχουμε καταφέρει σε λίγα χρόνια μονάχα να επιτύχουμε τόσα πολλά. Ήμασταν 21η από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Τώρα είμαστε η δεύτερη χώρα σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Έχουμε μειώσει το εθνικό χρέος από 85 σε 75% του ΑΕΠ και έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την αργία από το 11% στο 7% και ελπίζουμε ότι σε λίγα χρόνια θα είμαστε στην πλήρη απασχόληση. Κυρίε και κύριοι όμως δεν είναι αυτό το οποίο θέλετε εσείς να συζητήσετε από ό,τι κατάλαβα. <clears throat> θέλετε να μιλήσετε για την κατάσταση στην Ουγγαρία σε ό,τι αφορά πολιτικά ζητήματα και θέματα μετανάστευση. Για τα πολιτικά αυτά ζητήματα μπορώ να σας πληροφορήσω η Ουγγαρία είναι το κράτος μέλος το οποίο έχει εξεταστεί τις περισσότερες φορές από όλες τις φορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την ισχύ του κράτους δικαίου τα θέματα δημόσιας τάξης, τα θέματα μετανάστευσης, το κράτος δικαίου. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα, είναι θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλους μας. Είτε έχουμε τις σωστές ή όχι αποφάσεις για αυτό το θέμα, αυτό θα προσδιορίσει και τη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Πού μπαίνει τώρα η Ουγγαρία σε αυτό το θέμα. Οι Ούγγροι είναι σαφείς και αντιμετωπίζουν κατά πρόσωπο δύσκολες ερωτήσεις, δύσκολα προβλήματα. Δεν θέλουμε να μιλάμε με περιστροφές, αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα θέματα όπως η θανατική ποινή, όπως η μετανάστευση. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε μονάχα πολιτικά ορθές συζητήσεις, γιατί δεν μας έχουν φέρει πιο κοντά σε οποιαδήποτε λύση οι πολιτικά ορθές συζητήσεις. Πρέπει να μιλήσουμε ειλικρινά <clears throat> και ανοιχτά για το γεγονός ότι εμείς οι Ούγγροι Θέλουμε η Ευρώπη να είναι η Ήπειρος των Ευρωπαίων και θέλουμε η Ουγγαρία να ανήκει στους Ούγγρους. Όλα αυτά είναι, πιστεύω, απόλυτα συμβατά με τις ευρωπαϊκές αρχές και τις αρχικές ιδέες των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων και της μετανάστευσης από έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ μεταναστών και ετούντων άσυλο. Υπάρχουν οι οικονομικοί μετανάστες που απλώς ψάχνουν να βρουν μια καλύτερη ζωή. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, κύριε Τίμερμανς, δυστυχώς στην Ουγγαρία δεν μπορούμε να δώσουμε θέσεις εργασίας σε όλους αυτούς τους μετανάστες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά πρόσωπο και με ειλικρίνεια. Η οικονομική μετανάστευση είναι ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και η Ουγγαρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα της οικονομικής μετανάστευσης. Είμαι πεπισμένο λοιπόν ότι η πρόταση η οποία έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απλά λόγια είναι παράλογη και πλησιάζει τον παραλογισμό. Είναι πάρα πολύ λανθασμένο για μας να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, σαν ανοίξουμε τις πύλες της Ευρώπης, σας έρθει όποιος θέλει. Δείτε τα γεγονότα από μόνα τους. Είναι μια μεγάλη πρόκληση η μετανάστευση. Έναντι του 2010 έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των μεταναστών στην Ευρώπη μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αν δείτε και τις παράνομες διελεύσεις συνόρων, έχει 20 πλασιαστεί ο αριθμός των μεταναστών που έρχονται. Πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για το θέμα αυτό. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τους τωρινούς κανόνες, τις τωρινές συμφωνίες και τα κράτη-μέλη της Ευρώπης θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προστατεύσουν τα σύνορά τους. Αυτό είναι μια πραγματιστική και βιώσιμη λύση στα προβλήματα αυτά. Είναι <clears throat> παραλογισμός να προτείνουμε να μπουν όλοι οι μετανάστες στην Ευρώπη και να εφαρμόσουμε μονάχα τεχνητές ποσοστώσεις για να τους διανύμουμε στα κράτη-μέλη. Οι ποσοστώσεις το μόνο που θα κάνουν είναι να προσελκύσουν περισσότερους μετανάστες στην Ευρώπη. Είναι ένα κίνητρο για τους διακινητές και θα, ουσιαστικά θα παροτρύνουν τα, τους μετανάστες να διασχίσουν τη Μεσόγειο όσο επικίνδυνο και να είναι. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν που πιστεύω πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Εγώ χαίρομαι που επιτέλου συζητούμε αυτό το πρόβλημα. Αντί για ένα σύστημα ωστόσο, θα πρέπει κάθε μεμονωμένο κράτο μέλο να αποφασίσει για τον εαυτό του. Οι Ούγγροι θέλουν να αποφασίσουν από μόνοι του αν θέλουν μετανάστε ή όχι. Είμαστε μια χριστιανική κυβέρνηση και οι πραγματικοί αιτούντες άσυλο θα γίνουν δεκτοί, αλλά όχι όλοι οι οικονομικοί μετανάστες, γιατί δεν είναι ετούντε ασύλου, είναι απλώς άτομα τα οποία ψάχνουν για μια καλύτερη ζωή. Η παράνομη διέλευση των συνόρων είναι ένα δίκημα και πρέπει να δράσουμε εναντίον του. Η Ουγγαρία πρέπει να προστατεύσει τα σύνορά τη το κράτο δικαίου. Δεν θέλουμε να γίνουμε μια χώρα προορισμού για του παράνομού μετανάστες. Κάποιε χώρε μπορεί να θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό το σεβόμαστε πλήρω. Αλλά γι' αυτό το λόγο εμεί κάναμε αυτή τη δημόσια διαβούλευση για τα θέματα τη μετανάστευση. Νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό να ζητήσουμε από το λαό μα να αποφανθεί για το θέμα αυτό. <coughs> Είπε κάποιο βουλευτή ότι δεν πρέπει να γίνει δημόσια διαβούλευση για τη θανατική ποινή. Όχι, αυτό είναι μια παρεξήγηση. Δεν υπήρξε καμία δημόσια διαβούλευση για τη θανατική ποινή στην Ουγγαρία. Η Ουγγαρία δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία για το τι μπορούμε ή δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Και δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο κράτος μέλος έχει υπογράψει μια συμφωνία αυτού του είδους ή μια συμφωνία για το τι μπορεί να είναι αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης. Δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, δεν υπάρχει καμία τέτοια ε, επιταγή. Η συνθήκη προσχώρησης Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέει πουθενά για τι θέμα μπορούμε να συζητήσουμε και τι είναι ταμπού. Πιστεύω λοιπόν ότι οποιοδήποτε ο οποίος προσπαθεί να μας πει τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως Ούγγροι, τι πρέπει να συζητάμε, αυτό αποτελεί μια παραβίαση των ίδιων των συνθηκών. Αν δείτε τον αριθμό των αιτήσεων ασύλου που αντιμετωπίζει η Ουγγαρία, η δεύτερη με κριτήριο το ΑΕΠ της είναι η δεύτερη χώρα <clears throat> σε αριθμό αιτήσεων. Αν συγκρίνουμε τον αριθμό των αιτήσεων στον αριθμό των ε, πολιτών, είμαστε η 12η χώρα μετά από την ε, Σουηδία. Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα των Δυτικών Βαλκανίων. 43.000 αιτήσει έγιναν στο πρώτο μισό του 2014 ε, και οι μισές από αυτές περίπου από Κοσοβάρους. Είναι φανερό ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία με άτομα τα οποία ε, έρχονται από τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να θυμηθούμε ότι υπάρχει και η πρόκληση της Ουκρανίας. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της θανατικής ποινή. δεν μπορούμε να βάζουμε το κεφάλι, δεν μπορούμε να βάζουμε το κεφάλι μας <clears throat> στην ε, άμμο. Δεν είμαστε στο μεσαίωνα που δεν μπορούμε να μιλάμε για ορισμένα θέματα. Αυτό δεν αφορά συγκεκριμένα την θανατική ποινή, είναι θέμα ελευθερίας σκέψης και ελευθερίας έκφρασης θα πρέπει να μπορούμε να μιλήσουμε και για τη θανατική ποινή. Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να συνάδει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και το Σύνταγμα της Ουγγαρίας. Δεν είναι όλα αμετακίνητα και χαραγμένα σε πέτρα. Όλοι αυτοί οι κανόνες που ισχύουν έχουν δημιουργηθεί από τους ανθρώπους και μπορούν να αλλάξουν από τους ανθρώπους. Αυτή είναι η ελευθερία, αυτή είναι η δημοκρατία κυρίες και κύριοι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ό,τι πιστεύει. Μπορείτε να είστε επίτροπος, φιλόσοφος, πρόεδρος μιας πολιτικής ομάδας, αλλά η άποψή σας είναι η άποψη ενός πολίτη. Δεν υπάρχει μια ε, αλήθεια εκ των άνω, μια θεϊκή αλήθεια. Γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε την ελευθερία και αγωνιζόμαστε για την ευρωπαϊκή αξία της ελεύθερης σκέψης και της ελεύθερης έκφρασης ganz sicher gibt es keine göttlichen gebote die Σίγουρα δεν υπάρχουν θεϊκές επιταγές στις ευρωπαϊκές ε, συνθήκες, αλλά υπάρχει μια ανθρώπινη επιταγή, ου φωνεύσεις, λέει ο πρόεδρος Σούλτς. Ο κύριος Κονσάλες Πόνς για το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Κάποιες ομάδες θέλησαν να ξεκινήσουν στο σώμα μια συζήτηση για την Ουγγαρία. Εμεί δεν είμαστε αντίθετοι με τη συζήτηση οποιοδήποτε θέματος στο Κοινοβούλιο. Αυτό που δεν μας βρίσκει σύμφωνου είναι να κατηγορείται, να στιγματίζεται ένα κράτο μέλος τη Ένωση για πολιτικού λόγου. Επιτρέψτε μου να πω ότι καταρχά για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα η θανατική ποινή είναι ένα θέμα που δεν πρέπει ποτέ να επανέλθει στη συζήτηση. Είναι ένα σαφέ ξεκάθαρο θέμα αποφασισμένο, όπως η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όλοι οι Ευρωπαίοι ξεπεράσαμε τα χειρότερε τις στιγμές του παρελθόντος μας. Επιτρέψτε μου να σας πω επίσης ότι δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η Ουγγαρία θα τηρεί το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει ρητά την θανατική ποινή και καταδίκη. Και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό κ. Όρμπαν που ήρθε εδώ, που μίλησε μπροστά στο Κοινοβούλιο υποστηρίζοντας τις θέσεις του ενώπιον όλων ημών. Κυρίε και κύριοι, η μετανάστευση είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι επίση ένα πρόβλημα όπου οι πολιτικοί θα πρέπει να το βλέπουμε με μεγάλη προσοχή. Διότι όλοι είμαστε κατά της ξεφωνοφοβίας και του ρατσισμού και της ενοχοποίησης των Βρυξελών ταυτόχρονα. Η Ουγγαρία δεν είναι η μόνη χώρα όπου ε, αυξάνεται ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Σε όλη την Ευρώπη αυξάνονται. Δεν είναι η μόνη χώρα η Ουγγαρία όπου αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός, αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη. Θα κάναμε λάθος αν θεωρούσαμε ένα, ως ουγγρικό πρόβλημα ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Διότι πολιτικοί λόγοι κατά των μεταναστών, πολιτικοί λόγοι κατά της Ευρώπης γίνονται στη Γαλλία, την Ισπανία, την Γερμανία, τη Βρετανία, όλη την Ευρώπη. Δεν συζητούμε την, ενοχή της Ουγγαρίας, αλλά τη δική μας ενοχή για την ανικανότητά μας να μπορέσουμε να κάνουμε σεβαστές τις αξίες της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού εγχείρημα παντού. Αυτό δεν έγινε για να δικάσουμε οποιοδήποτε κράτος. Αν το κάνουμε αυτό εδώ μπορεί και εμείς να κάνουμε όπως ε, αυτά που θα κινδυνεύσουν να κλονίσουν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Κονσάλε Πόνς. Για τη σοσιαλιστική ομάδα έχει ο κύριο Νίτερ Μίλλερ τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως σας φαίνεται παράξενο, αλλά εγώ πρέπει να πω ότι δεν χαίρομαι που είναι παρόν ο Πρωθυπουργό τη Ουγγαρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί, γιατί κάθε φορά που έρχεται εδώ πέρα τα πέντε πέντε αυτές φορές που έχει έρθει έχουμε μιλήσει για την επονίδιστη πολιτική της κυβέρνησής μας και αυτές οι συζητήσεις σπηλώνουν τη χώρα μου. Εγώ θα πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι ξενόφοβη η Ουγγαρία. Η χώρα μου δεν είναι κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας πάντα στρέφεται κατά των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι οι αρχές επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάει για αυτό, αυταρχικές πολιτικές, για ανελεύθερη δημοκρατία, την επιτυχία των αυταρχικών συστημάτων. Συζητήσεις όπου η δημοκρατία θεωρείται ότι είναι μια ανοησία. Αυτό το έχει πει ο Πρωθυπουργός μας. Ναι. Υπάρχουν ε, παραπληροφορήσεις στους... Ε, παραπληροφορούνται οι Ούγγροι και ουσιαστικά παροτρύνονται να έχουν μια στάση μίσους, γιατί η κυβέρνηση πάει να ψαρέψει τις ψήφους των ε, ακροδεξιών κομμάτων, επειδή χάνουν ψηφοφόρους. Προσπαθούν να βρουν νέους ακροδεξιούς υποστηρικτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν μπορεί να δεχτεί αυτές τις πολιτικές Δεν είναι μονάχα ε, δεν η Ουγγαρία η οποία φταίει όλα αυτά, αλλά η δράση της τωρινής Ουγγρικής κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο για την ομάδα των φιλελευθέρων στον πρόεδρο Φερχόφστατ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν από τους πρώτους που ήθελα να ακούσω τον κύριο Ορμπάν, αλλά αυτά που ήρθε να κάνει εδώ είναι απλώς να συνεχίσει τις προκλήσεις που ακούσαμε και τον περασμένο μήνα στην Ουγγαρία και εκτός αυτής. Δηλαδή, στη μέση της κρίσης με την Ουκρανία συνήψε ενεργειακή συμφωνία με τον κύριο Πούτιν και μετά η θανατική ποινή, άλλη πρόκληση. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε απόψεις κύριε Ούρμπαν. Την 1η Μαΐου, την Πρωτομαγιά είπατε στο δημόσιο ραδιόφωνο στην Ουγγαρία ότι αυτό που θέλετε είναι κάθε χώρα μέλος να μπορεί να αποφασίζει μόνη της για την επαναφορά της θανατικής ποινής, ότι δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα και το επιβεβαιώσατε και σήμερα, ενώ είναι ευρωπαϊκό θέμα. Δεν είναι θέμα κράτους, είναι θέμα ολόκληρης της Ένωσης και του ολόκληρου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Τέλος, και πάλι το επιβεβαιώσατε, άλλη πρόκληση, είπατε κάνω μια εθνική διαβούλευση απλώς για τις μεταναστεύσεις. εθνική διαβούλευση είναι αυτή. Διαβάστε, διαβάστε εδώ τα ερωτήματα που τίθενται. 7. Έβδομο ερώτημα. Υποστηρίζετε την κυβέρνηση για πιο αυστηρή νομοθεσία για τους μετανάστες αντίθετα με την πολιτική των Βρυξελών. Άρα οι Βρυξέλλες φταίνε. Ερώτηση 3. Απίστευτη. Απίστευτη. Μερικοί θεωρούν ότι η κακοδιαχείριση του μεταναστευτικού από τις Βρυξέλλες μπορεί να έχει κάποια σχέση με την αύξηση της τρομοκρατίας. Η Ευρώπη και οι Βρυξέλλες δηλαδή ευθύνονται για την αύξηση της τρομοκρατίας και το ξαναείπατε πάλι. Αυτό είναι εθνική διαβούλευση. Εγώ το λέω ρητορικά ερωτήματα γιατί έχετε ήδη την απάντηση. Δεν χρειάζεται να δοθεί άλλη. Τέλος, σκεφτείτε ένα πράγμα. Αν επιτίθεστε κατά των μεταναστών, σκεφτείτε τους Ούγκρους πρόσφυγες που άφησαν τη χώρα τους λόγω του κομμουνιστικού καθεστώτος από το 1956 και μετά και πώς έγιναν δεκτοί με ανοιχτές αγκάλες από άλλους λαούς της Ευρώπης. Για τους πράσινους η κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο. Μια στιγμή κυρία Σαρτζεντίνη. Είχα πει πριν από αυτό το γύρο δεν θα υπάρξουν μπλε κάρτες. Ίσως ε, ε, ήσασταν απόν και δεν το καταλάβατε. Κυρία Σαρτζεντίνη, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, τα λόγια μπορεί να είναι λουλούδια, αλλά μπορεί να είναι και στιλέτα. Εμείς παίζουμε με τις λέξεις και οι λέξεις, ε, οι λέξεις κύριε Όρμπαν δεν είναι πέταλα, είναι σφαίρες. Έχει κανείς την εντύπωση ότι μπορεί να είναι πέταλα λουλουδιών, αλλά τα λόγια που χρησιμοποιείται ε, λειτουργούν ως όπλα. Και δεν μιλάμε μόνο για λόγια, μιλάμε και για πράξεις όταν μιλούμε για τη θανατική ποινή, όταν μιλούμε για το ότι ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε τη διαβούλευση αυτή με την εξαιρετικά μεροληπτική διαβούλευση ως ένα απλό γεγονό. Έρχεστε και μας λέτε τι γίνεται με τη μετανάστευση και το πρόγραμμα της Επιτροπής, ενώ λέτε ότι δεν πρέπει να ανοίγουμε τις τρόφιγγες. Αυτό είναι το ζήτημα η ανευθυνότητα ενός πρωθυπουργού μιας χώρας. Αυτή η ευθύνη είναι μια ευθύνη δική σας και ευθύνη που σας δεσμεύει. Ο κύριος Μάιερ από τις μια εγγεγραμμένος <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν κάνετε μια πολιτική δήλωση δεν πρέπει να την κάνετε ως πρόεδρος, θα πρέπει να την κάνετε από τα κάτω έδρα της Ολομέλειας. Ένα, ένα πράγμα θέλω να πω από την αρχή για μας υπάρχει αναμφισβήτητα η απαγόρευση θανατικής ποινής. Αλλά υπάρχει το δικαίωμα να συζητήσει για κάτι τέτοιο. Εμείς συζητάμε για κάτι το οποίο είναι υποθετικό και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ιστερική η αντίδραση των αριστερών. Και από τη δική τους πλευρά πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό. Το γεγονός ότι μια δεξιά κυβέρνηση μπορεί να είναι επιτυχημένη και να έχει την υποστήριξη των πολιτών. Και γι' αυτό είναι αυτό το σκάνδαλο. Είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για τα θέματα αυτά της Ουγγαρίας και που υπάρχει αυτή η προσπάθεια παρέμβασης στα, στα εσωτερικά της. Η Ουγγαρία που είχε πολύ κακές εμπειρίες στο παρελθόν θα ήθελα να τους πω, άμα θέλετε να παρέμβετε, τότε να παρέμβετε στους συντρόφους σας, να πάτε στην Ελλάδα να παρέμβετε. Νομίζω ότι αυτό που έχει γίνει είναι απόλυτα λαθασμένο. Ευχαριστώ. Για την ομάδα του ΕΛΚΟ, κύριο Ζάιρ έχει το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, η συζήτηση αυτή ήταν, είναι όμοια με τις προηγούμενες μια συζήτηση μεταξύ κοφών. Ο ένας δεν ακούει τον άλλον. Ο κύριος Βεχόφστατ δεν ήθελε να ακούσει τα, το σχόλιο του κυρίου Όρμπαν ότι είμαστε δημοκράτες και ότι οι πόρτες Ουγγαρίας είναι ανοιχτέ σε αιτούντες άσυλο. Δεν θέλησε να ακούσει την δήλωση αυτή. Αναφέρθηκε στους, αναφερθήκατε στους πρόσφυγες του 56. Αυτό είναι μια χαμηλού επίπεδου πολιτικάντικη κουβέντα. Μιλήσατε για, διαβάσετε τα ερωτήματα της διαβούλευσης, κύριε Φερχόφσταντ. τον πολίτη της Ουγγαρίας για κάτι τόσο σημαντικό όπως θέλετε αυστηρότερους κανόνες, γιατί αυτό θεωρείτε ότι είναι αντιδημοκρατικό. Δεν πρέπει να περιμένεις απαντήσεις όταν θέτεις ερωτήματα είναι μια, ένας διάλογος κοφών και το μόνο στο οποίο μας οδηγεί είναι σε αδιέξοδο. Καταλαβαίνω ότι ως πρώην απικιακές δυνάμεις βιώνεται μια διαφορετική κουλτούρα στην υποδοχή μεταναστών από άλλες χώρες. Εμείς δεν είμαστε ε, απικιακή δύναμη παλιά. Δεν έχουμε συνηθίσει τους μετανάστες. Δεν ξέρετε τι σημαίνει να εμφανίζονται στα σύνορά σε χιλιάδες άνθρωποι και να μην μπορεί να διακρίνει αν είναι οικονομικοί μετανάστες ή ετούντες άσυλο. Η Ουγγαρία είναι η δεύτερη χώρα μετά τη Σουηδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αιτήσεων ασύλου. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία σας στην διαμόρφωση της πολιτικής. Βλέπω ότι κουνάει το κεφάλι σας. Τι είπα λάθος. Πριν από 20-30 χρόνια κάνετε λάθος πολιτική. Λάβατε μια λάθος απόφαση πολιτικής στη μετανάστευση. Πρέπει να είμα... Εμείς θέλουμε να μην το κάνουμε αυτό το λάθος. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί για να αποφύγουμε την ξενοφοβία. Η, η ειρηνική συνύπαρξη είναι βασικό ζήτημα στην Ευρώπη. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για αυτή την ελληνική συνύπαρξη. Ο κύριος Βάιντεν Χόλτζερ για τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι είναι ήδη αμφισβητήσιμο το γεγονός ότι έπρεπε να έρθετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είσαστε μαέστρος ικανός στο να έχετε διπλή γλώσσα και στην ασάφεια καταφέρετε, καταφέρετε πολύ καλά. Το ερώτημα είναι ποια είναι η απόψή σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνετε για να αντιμετωπίσετε την τρομερή διαφθορά που υπάρχει στη χώρα σας. Τι έχετε κάνει για να αντιμετωπίσετε το γεγονός ότι τόσο πολλοί Ούγγροι χρειάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τους και να εργαστούν εκεί τι έχετε κάνει για να δημιουργήσετε ένα κλίμα συμφιλίωσης στη χώρα σας. Αυτά τα ερωτήματα τα θέτουμε ως φίλοι της Ουγγαρίας και επειδή γνωρίζουμε όλη τη σημαντική συνεισφορά του λαού της Ουγγαρίας για την επίτευξη της δημοκρατίας και της ελευθερίας στην Ευρώπη. Για τους φιλελεύθερους ο κύριος Μισελ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Κύριε Ορμπάν, λέτε ότι σας αρέσει η ειλικρίνεια. Πολύ ωραία. Θα σας μιλήσω λοιπόν και εγώ ειλικρινά. Κύριε Ορμπάν, οδηγείτε τη χώρα σας σε μια αυταρχική οδό που δεν συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές ουμανιστικές ανθρωπιστικές αρχές. Η αριθμητική είναι μέρος της δημοκρατίας αλλά δεν αρκεί. Στην πραγματικότητα κάνετε αυτό που ονομάζουμε τυραννία της πλειοψηφίας. Έχετε πλειοψηφία και νομίζετε ότι έχετε το δικαίωμα έτσι να κάνετε ό,τι θέλετε και να καταπιέζετε τις μειονότητες και τους ε, αντιφρονούντες. Μιλάτε για τη θανατική ποινή, το ερωτηματολόγιο σας ε, είναι ρητορικά τα ερωτήματά του και τελικά όλα αυτά δείχνουν μεθόδους που αντιτίθενται πλήρως στο πνεύμα και το γράμμα των συνθήκων πονηρά και δημαγωγικά καταχράστε την ίδια την ιδέα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ενθαρρύνετε το ρατσισμό και τη ξενοφοβία και τη μυσαλλοδοξία. Μιλάτε για ρίζες και μειώνετε την ελευθεροτυπία και την ανεξαρτησία του δικαστικών αρχών και επίσης εκφοβίζεται τον κόσμο. Σιγά σιγά δηλαδή με σιγανή φωτιά καίτε όλες μας τις αξίες και παραβιάζεται τις ιερότερες αρχές της Ένωσης και του κράτους δικαίου. Ένα καταπληκτικό λαό τον οδηγείται σε ορμή αντίθετη από τις ιστορίες προς τον ολοκληρωτισμό. Πώς ακόμη θα ανεχτούμε πλέον εμείς οι ανθρωπιστέ κύριε Τίμερμανς από αυτό το καθεστώς που κοινικά μιλάει για τον εαυτό του και μόνο και να οδηγήσει σε απόλυτο καθεστώς, σε απόλυτη εξουσία. Το, τον λόγο τώρα για τους πράσινους έχει κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κύριοι Πρωθυπουργέ. Το θέμα εδώ πέρα δεν είναι δεξιά-αριστερά, είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες. Και θα πρέπει να έχουμε την ίδια στάση ανεξαρτήτως κόμματος. Ως πράσινη δε εμείς πούμε κριτική και στη δική μας κυβέρνηση. Πρόκειται για τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναφερθώ για το ερωτηματολόγιο της ε, μετανάστευσης ε, που στείλατε στους πολίτες σας που προωθεί τις προκαταλήψεις. Ο κύριος Βέμπερ και εσείς μιλήσατε για τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της χώρας σας. Αλλά τότε γιατί έφυγαν 500.000 άνθρωποι από τη χώρα σας τα τελευταία χρόνια για να βρούνε δουλειά ή καλύτερη ζωή σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτός είναι ο ε, διπλάσιος αριθμός από όσους έφυγαν από τη δικτατορία του 56. Γιατί εμποδίζετε τους φοιτητές να φύγουν από τη χώρα και τους λέτε πως πρέπει να πληρώσουν τα δίδακτρα εάν δεν μείνουν στη χώρα. Μήπως θα πρέπει να κάνετε ένα ερωτηματολόγιο για να δείτε πώς μπορείτε να κρατήσετε τον κόσμο στη χώρα σας αντί να σηκώνετε να φεύγει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόγκορ τώρα για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προασπίσουμε τα ευρωπαϊκά μας κεκτημένα. Ταυτόχρονα όμως είναι εξίσου σημαντικό να προστατεύσουμε και τις παλιές ευρωπαϊκές παραδόσεις όπως την ελεύθερη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζήλευτη ανά τον κόσμο γιατί ακριβώς ε, μπορούμε να συζητάμε με διαφορετικές απόψεις με βάση αντικειμενικά γεγονότα. Και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και προσπαθούμε να πείσουμε ο ένας τον άλλον. Είμαι λοιπόν πεπισμένος πως πρέπει να διατηρήσουμε αυτές τις αξίες. Γι' αυτό θα ήθελα να συζητάμε σοβαρά κάποια ζητήματα και όχι μόνο για να επιτύχουμε κάποιες πολιτικές νίκες. Συνεχώς κάποιες κυβερνήσεις είναι στο εδόλιο. Η κυρία Λούνατσεκ μας είπε για 3 εκατομμύρια ανθρώπους που έφυγαν, έφυγαν από τη Ρουμανία 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Ε, δεν ε, συζητάμε όμως ποτέ τη Ρουμανία για την δε Σλοβακία και τα διατάγματα Μπένες ε, και τα διατάγματα περί Εκεί πέρα δεν λέτε τίποτα γιατί είναι σοσιαλιστές. Ευχαριστώ για τους ε, σοσιαλδημοκράτες ο κύριος Ουέλη. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι Ούγγρος ε, και σοσιαλδημοκράτης ε, Ευρωπαίος. Γι' αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω πως η Ουγγαρία την οποία περιγράφει ο κύριος Όρμπαν δεν είναι η Ουγγαρία, είναι ένα έσχος. Η εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση Όρμπαν είναι έσχος και θέλω να πω πως η Ουγγαρία έχει και άλλη μια όψη. Τούτου λεχθέντος. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός δεν ανησυχεί τόσο πολύ για τη θανατική ποινή, τη μετανάστευση, τη διαβούλευση. Όχι, τον ενδιαφέρουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο που στηρίζουν ένα σύστημα στη χώρα μας ε, το οποίο χρησιμοποιεί για να κατευθύνει τον Ουγγρικό λαό. Οπότε μην μιλάτε εξ ονοματός μου κύριε Πρωθυπουργέ και εξ ονόματος των εκατοντάδων χιλιάδων που έφυγαν από τη χώρα και μη μιλάτε εξ ονόματος ε, όσων μου έστειλαν αυτό το ρετματολόγιο για να το σκίσω μπροστά σας. Γιατί αυτό είναι πρόκληση. Ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους, κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ πολύ. Για πόσο χρόνο ακόμα θα συνεχίσει η κυβέρνηση του κυρίου Όρμπα να σοκάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από μια σειρά δράσεων και προτάσεων οι οποίες αποτελούν διακριτική μεταχείριση και μας οδηγούν και πάλι να συζητάμε σήμερα την Ουγγαρία. Σας ρωτώ κύριε Όρμπαν, αυτό σας χαροποιεί, σας αρέσει να είστε προκλητικός, θέλετε εσείς να αμφισβητείτε τις αξίες πάνω στις οποίες χτίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα μιλήσατε για την θανατική ποινή ε, και την επανεισαγωγή αυτή. Στείλατε ένα ερωτηματολόγιο στους πολίτες σας. Αυτό είναι πρόκληση απλά. Είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Ούγγροι και σας διαβεβαιώ πως πολλά τα μέλη του, του Κοινοβουλίου που θα κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν διασφαλίσουν τα βασικά τους δικαιώματα. Ακόμα και αν εσείς και η κυβέρνησή σας κύριε Όρμπαν κάνετε ό,τι μπορείτε για να υποσκάψετε τα δικαιώματα αυτά. Εάν μου επιτρέπετε λοιπόν θα ήθελα να διαβάσετε το Σάντορ Μάρε που είναι ένας από τους μεγάλους Ούγγρους συγγραφείς του 19ου αιώνα. Ούγγρος λοιπόν και αυτός και αν ήταν σήμερα εν ζωή θα έχει λογοκριθεί από εσάς ίσως θα έπρεπε να αποτελέσει ένα ηθικό παράδειγμα για να ακολουθήσετε, γιατί μιλά για τα βασικά δικαιώματα και αξίες κάθε ατόμου. Ε, θα Έπρεπε λοιπόν για σας να αποτελεί ένα παράδειγμα που να ακολουθήσετε και εσείς και η κυβέρνησή σας. Ο κύριος Γιάβορο για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σα υπογραμμίσω πως έχουμε κάποιες κοινέ ευρωπαϊκές αξίες και για να πείσετε τους εταίρους σα ήρθατε εδώ και μας είπατε πως το ΦΙΝΤΕΣ αποτελεί το θέμα το φύλακα που ε, ουσιαστικά εμποδίζει την άκρα δεξιά από το να κερδίσει και άλλο έδαφος. Ίσως παρατηρήσατε πως όλο και συχνότερα πλησιάζετε τις θέσεις της άκρας ε, δεξιάς. Μιλάμε για πολιτικό έδαφος το οποίο ψάχνετε να κερδίσετε και η σημερινή πολιτική συζήτηση ε, δείχνει πως και εσείς κύριε Βέμπερ θα πρέπει να δεχτείτε την πραγματικότητα. Η στρατηγική αυτή δεν έχει πετύχει. Έχουμε κάποιες ριζοσπαστικές ε, δηλώσεις από πλευρά σας που δεν σας βοήθησαν να κερδίσετε ψήφους. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι σας απλώς συνήθισαν ένα επίπεδο συζήτησης το οποίο στο παρελθόν ε, στήριζε μόνο άκρα δεξιά. Το μόνο το οποίο θεωρώ ότι στη δική σας κυβέρνηση είναι ε, συνεπές είναι ότι έχετε διαφθορά και πολλά προβλήματα στη χώρα σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως εσείς είστε στην αιχμή του δόρατος στην Ουγγαρία και βοηθάτε εσείς τη χώρα σας να σταθεί στα πόδια σας ή θα σας θυμούνται για κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ για το ΕΛΚ ε, τώρα κυρία Γκάλ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρίμα κύριε Πρόεδρε που δεν μας επιτρέψατε να κάνουμε ερωτήσεις γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Πρώτα απ' όλα διαβούλευση για τη θανατική ποινή. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια διαβούλευση. Κύριε Φερχόφστατ, για τους πρόσφυγες. Τους καλωσορίζουμε να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ ε, παρανόμων οικονομικών μεταναστών και προσφύγων. Αυτά για τον κύριο Φερχόφστατ. Τώρα, για την ε, ελευθερία ε, μετακίνησης, ε, αυτό είναι και εκτιμένο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινό για όλους. Ε, γιατί ασκείται κριτική στον Πρωθυπουργό μας όταν ο κόσμος εξασκεί ένα δικαίωμα, ένα δικαίωμά του. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί μας κρίνεται σε ένα ηθικό επίπεδο, κυρία Βίξτρομ, ποιος σας όρισε κριτή. Και επιπλέον για την κατάσταση. Ε, είχαμε οικοσαπλασιασμό των ανθρώπων που εισέρχονται στην ε, χώρα μας. Οπότε λογικό είναι να υπάρχει κάποια αναστάτωση. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πώς ε, ζει ο κόσμος αυτό το φαινόμενο. Και με κάθε ερώτηση έχουμε συμφωνείτε, διαφωνείτε και ο καθένας μπορεί να απαντήσει. Ο κάθε πολίτης απαντά αν συμφωνεί ή όχι. Για μας αυτό είναι η δημοκρατική διαδικασία. Τώρα, πράγματι, ε, δεν τα κάνουμε σύμφωνα με τον ευγενικό τρόπο των διαδρόμων των Βρυξελών. Θέλουμε να μάθουμε τι λέει ο πραγματικός κόσμος. Υπήρξε μια επιστολή που υπέγραψαν εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγροι πολίτες και είναι κρίμα που δεν αναγνωστεί γιατί οι περισσότεροι Ούγγροι θεωρούν πως είναι άχρηστη η συζήτηση. Ευχαριστώ για τους σοσιαλδημοκράτες. Η κυρία, ε, ο κύριος Σίλβα Περέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς ο κύριος Όρμπερν δεν ήρθε εδώ ε, για να μας δώσει διευκρινήσεις ε, ούτε και για να επαναβεβαιώσει την πίστη του προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και προς τις ε, βασικές δημοκρατικές αρχές απλώς ακούμε διάφορες ε, απειλές ε, ε, εναντίον όσων ασχολούνται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το χειρότερο δε είναι ότι αυτό το πράττει με την βοήθεια και την συνενοχή διαφόρων βουλευτών του και του δικού μας Κοινοβουλίου και από το ΕΛΚ. Αυτά τα θέματα θέματα βεβαίως μπορείτε να τα συζητάτε στην Ουγγαρία όσο θέλετε αλλά ε, εάν ε, κάνετε τέτοιου είδους πράξεις και παίρνετε τέτοιες αποφάσεις τότε θα πρέπει να περιμένετε ε, οτιδήποτε περιμένει αυτούς που αντιτίθενται και παραβιάζουν τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις δημοκρατικές αρχές. Περνάμε τώρα στη διαδικασία. ΚΕΤΣ Η κυρία Πίτυρ. Ευχαριστώ πολύ. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η προώθηση των ανθρωπίνων αξιών αποτελεί προτεραιότητα της Ουγγρικής κυβέρνησης και αποτελεί και τμήμα των συνταγματικών δικαιωμάτων της χώρας. μιλήστε για να δω εάν υπάρχει διερμηνία, αλλά πρέπει να, να πείτε κάτι για να μεταφραστεί. Αν δεν λέτε τίποτα, δεν ακούω κι εγώ τίποτα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προώθηση των ανθρωπίνων αξιών είναι πολιτική της Ουγγρικής κυβέρνησης και τμήμα των συνταγματικών δικαιωμάτων στη χώρα. Οι αρχές αυτές και οι αξίες που ακολουθούν είναι διαφορετικές από τις δικές μου. Και πρέπει να σας πω πως διάβασα τη δήλωση του κυρίου Όρμπαν και δεν βρήκα πουθενά ε, να δηλώνει κάτι για το οποίο έχει κατηγορηθεί. Πιστεύω λοιπόν πως όσοι δεν μπορούν να κερδίσουν στις εκλογικές μάχες των Βίκτορ Όρμπαν με τον τρόπο αυτό αποδεικνύουν πόσο αδύναμη είναι. Ο Βίκτορ Όρμπαν προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών του. Δεν έχω δει να έχει κάνει καμία δήλωση κατά των προσφύγων και των ετούντων άσυλο. Το μόνο που ζήτησε είναι τη γνώμη των πολιτών του ε, για το πώς αντιμετωπίζουν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση. Δεν θεωρώ πως η Ουγγαρία θα πρέπει να καταδικαστεί για το γεγονός ότι ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Πιστεύω δε πως και άλλοι πολλοί πρωθυπουργοί οι οποίοι προέρχονται από ε, τους σοσιαλιστές θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του και κυρίως εάν δεν θέλουν να κάνουν δημοψήφισμα ε, να προσέξουν γιατί πολλές φορές ακόμα και το 1 τρίτο των πολιτών το ζητάει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος ε, Τσάλα. Περιμένετε λίγο. Τον συνάδελφο Τσάλα έδωσα τον λόγο, κύριε Τσάρνη, με συγχωρείτε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε την ε, συζήτηση. Ο κύριος ε, Βέμπερ προσπάθησε να αιτιολογήσει την αντιδημοκρατική συμπεριφορά λέγοντας ότι ε, υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή σαν να λέμε ότι δεν πειράζει η παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Κίνα γιατί και εκεί υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Για την κυβέρνηση του κυρίου Όρμπαν είδαμε πώς ε, γίνεται κατάχρηση της πλειοψηφίας, ε, πώς οι μειονότητες καταπιέζονται. Είστε ένα είδος Πούτιν που χρησιμοποιεί τις μειονότητες ε, και κατέληξε να τις χρησιμοποιήσει και για να εισβάλλει σε γειτονικές χώρες. Δεν είναι σωστή διακυβέρνηση αυτή, κύριε Ορμπάν. Πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να συζητήσουμε το θέμα αυτό, γιατί δεν είναι ο σωστός τόπος, αλλά κύριε Πρόεδρε, Νομίζω ότι αναφερθήκατε και εσείς στο άρθρο 2, αλλά όχι με μεγάλη ακρίβεια, γιατί η πρώτη παράγραφος του άρθρου αυτού λέει το εξής. Μία από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής. Σεβασμός της ανθρώπινης ζωής. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει παραμεληθεί και έχει αμφισβητηθεί. Θυμόσαστε τι συνέβη όταν υπογράφηκαν οι συνθήκες της Ρώμης. Δεν υπήρχε καμία δημοκρατική ε, χώρα στην Ευρώπη που δεχόταν το δικαίωμα στην άμβλωση. Αν λοιπόν σας ανησυχούν τόσο πολλοί αποκλεισμοί και ε, αναφέρεστε τόσο συχνά στην άρθρο 7 των Ευρωπαϊκών ε, Συνθήκων, τότε ίσως θα έπρεπε να αναρωτηθείτε και για τη δική σας θέση. Κυρία Πάγκα Όλη μας τη ζωή ψάχνουμε να δώσουμε απαντήσεις στα, στα σημαντικά ερωτήματα. Ο Σάντορ Μαρέι, ο μεγάλος Ούγγρος συγγραφέας, το είπε αυτό. Ήταν κατά του ναζισμού, ήταν κατά του φασισμού, ήταν κατά του κομμουνισμού, ανθρωπιστής, φιλελεύθερος, που έσκασε από την Ουγγαρία και βρήκε καταφύγιο στη ΣΥΠΑ. Νομίζω ότι σήμερα δεν θα μπορούσε καν να αντέξει την Ουγγαρία του Ορμπάν. Το να ζητήσει κανεί αν υπάρχει σχέση με την αύξηση τρομοκρατία και τη μεταναστική πολιτική τη Ευρώπη είναι να απαντά κανεί με. Ε, ξενόφοβο τρόπο τις ε, σημερινές ε, προκλήσεις. Το να είναι κανείς ε, να απαντήσει κανείς με τα ε, λόγια του Ούγκρου συγγραφέα, τα οποία διάβαζα και με ανακούφιζαν όταν με κυνηγούσαν στη χώρα μου, τη χώρα των Βάσκων. Με τρομάζουν ε, αυτά που λέτε κύριε Όρμπαν και εσείς κύριε Βέμπερ θα πρέπει να είστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε με κάποια κόλπα να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τέτοια μεγάλα προβλήματα. Είσαστε ένα μεγάλο ε, ευρωπαϊκό κόμμα κύριε Βέμπερ. Μην ακολουθείτε τέτοιου Μαραγκάλ, έχει το λόγο, παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου. Σε, escuchar a todo el Με ακούτε τώρα, πολύ ωραία. Ωραία. Εάν είναι να ακούσουμε κάτι παρόμοια με λόγια με τα όσα ακούγαμε προηγουμένως από τον κύριο Όρμπαμ να σας πω πως μόνο ανησυχία μπορεί να μας δημιουργήσει. Κινδυνεύει η ελευθεροτυπία και η ελευθερία της έκφρασης από τη σύνδεση τρομοκρατίας και μετανάστευσης. Δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτές τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας επειδή πάει καλά η ουγγρική οικονομία τέτοιου είδους εκστρατείες που είναι καθαρά ξενοφοβικές ε, μοιάζουν με τα όσα λένε κάποιοι ε, του Λαϊκού Κόμματος στις ε, τοπικές εκλογές στη χώρα μου. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε ε, το θέμα της Ουγγαρίας όπως κάνουμε ε, οποδήποτε έχουμε μία ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Έχουμε την υποχρέωση, όχι το δικαίωμα μόνο να συζητάμε αυτές τις παραβιάσεις και εδώ και σε άλλα κράτη όταν κινδυνεύουν οι βασικές δημοκρατικές αξίες όπως, κάνουν, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ισπανία όπου έχουν περιοριστεί τα δικαιώματα αυτοδιάθεσης των πολιτών της Καταλωνίας. Ευχαριστώ κύριο Σκοβάο Ευχαριστώ, Πρόεδρε Σούλτς. Ο Όρμπαν και η κυβέρνησή του νομίζω ότι οδηγεί την ε, ε, Ουγγαρία, τη χώρα του, στην ε, απολυτοκρατία και στην οπισθοδρόμηση καταπιέζει και καταστέλει τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και σιγά σιγά αρχίζει και ξανασυζητάει για την ε, ε, ε, θανατική ποινή. Μετά τι θα γίνει, θα αρχίσει το κυνήγι των μαγισσών ή μήπως η ιερά εξέταση. Ένας ε, Ιταλός συνομιλικός μου, ο Αντρέα Τζουλιάνο, ε, του ε, απειλείται η ζωή του και μάλιστα ε, έχει μπει κεφαλική ανταμοιβή από τον Γιώπικ και φαίνεται ότι αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Ο Ανδρέα Τζουλιάνο ζει μια κατάσταση εκτός πραγματικότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ζητώ λοιπόν η κύριε Όρμπαν κάντε κάτι έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ζωή αυτού του νεαρού. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, τελείωσε η διαδικασία και έτσι και η συζήτηση. Κύριε Όρμπαν, θέλετε να ξαναμιλήσετε αν θέλετε. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω πως ε, σας ευχαριστώ για όσα ακούστηκαν από την Ιταλία, από τις σκανδιναβικές χώρες, την Γερμανία. Θα ήθελα να πω το εξής. Εγώ ποτέ δεν θα τολμούσα να μιλήσω έτσι για τις χώρες και τους λαούς σας. Μάλιστα να πω κάτι τώρα και παρακαλώ... Α, ναι, κύριε Όρμπαν, ξαναξεκινήστε από την αρχή γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με την ε, διερμηνία. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακούσαμε ε, ε, Γερμανούς, Ιταλούς, Ισπανούς, εκπροσώπους από τις βαλτικές χώρες. Δεν θα ε, μιλήσω για κανέναν προσωπικά με το όνομά του, αλλά πραγματικά θα ήθελα να πω ότι δεν θα τολμούσα να φερθώ άσχημα στους εκπροσώπους των χωρών αυτών και στους πολίτες των χωρών σας. Δεν θα το άντυχε η συνείδησή μου. Θα ήθελα λοιπόν να δραχθώ τη ευκαιρία έτσι ώστε να σας μιλήσω για την Ουγγαρία και την αξιοπρέπειά μα. Ε, όσον αφορά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχονται από την ε, Ουγγαρία, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό σήμερα, γιατί εγώ δεν θέλω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει ένα είδος ε, ε φόρουμ ενδοουγγρικών διαφορών. Δυστυχώ όμω, βλέπω Ούγγρου βουλευτές να επιτίθενται κατά τη ίδια ίδιες τους της χώρας ε, και ε, λένε ότι δεν θα πρέπει να στηρίζεται πλέον η Ουγγαρία γιατί δεν την αξίζει αυτή τη στήριξη και αυτή τη βοήθεια. Ας το παραβλέψω όμως. Αναφέρεστε στην ε, δημοκρατία, δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα τα στοιχεία, πάντως πρέπει να πω ότι η φιλελεύθερη οικονομία δεν λειτουργούσε πάντα. Το 8 είχαμε μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση. Βλέπω ε, ε, με χαρά ότι ε, πολλοί μεταξύ μόνοι έχετε διαβάσει το Σάντορ Μάντοι. Χαίρομαι γι' αυτό, αλλά βεβαίως θα πρέπει να ξέρετε και με ποιο τρόπο και κάτω από ποιες συνθήκες εργάστηκε και έγραψε αυτός ο μεγάλος συγγραφέας. Κύριε Μισελ, είμαστε σε μια χώρα η οποία λειτουργεί με εκλογές. Τρεις φορές κέρδισα τις εκλογές, τρεις φορές τις έχασα. Αυτό είναι απολύτω δημοκρατική λειτουργία, έχω την εντύπωση. Ε, επίσης, ε, κύριε Πρόεδρε των Φιλελευθέρων, θα ήθελα να απαντήσω και σε εσά. Κατανοώ ε, τα κίνητρά σα και κατανοώ την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, γιατί ε, ήταν πολύ μεγάλο κόμμα οι φιλελεύθεροι στην Ουγγαρία και έπαιξαν μεγάλο ρόλο μετά τον κομμουνισμό, αλλά τώρα έχουν εξαφανιστεί από την πολιτική σκηνή και κατανοώ ότι αυτό ενοχλεί τους φιλελεύθερους της Ευρώπης, αλλά δεν, ε, οφείλ, δεν ευθύνονται οι Ούγγροι γι' αυτό το λόγο και οι Ούγγροι ψηφοφόροι. Ε, όσον αφορά την ε, διαβούλευση τώρα, ίσως θα πρέπει να μάθετε και μερικά πράγματα. Ο πρόεδρος της φιλελεύθερης ομάδας δεν θεώρησε ότι εμείς θα έπρεπε να υποβάλουμε το ερώτημα στηρίζεται την Ουγγρική γραμμή σχετικά με το να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες από ό,τι Βρυξέλλες. Κοιτάξτε, εμείς δεν είχαμε τέτοια προβλήματα μέχρι πρόσφατα. Ε, η Ουγγαρία είχε τη δικιά της εθνική νομοθεσία και είχαμε την δυνατότητα να καλωσορίζουμε πρόσφυγες οι οποίοι έφταναν στα Ουγγρικά σύνορα και μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Όμως το 2002 ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρέωσε την Ουγγαρία να αλλάξει ε, τους κανόνες της και να δέχεται και οικονομικούς μετανάστες. Αν δεν είχε υποχρεωθεί από την Ευρώπη η Ουγγαρία να τροποποιήσει την νομοθεσία της και τον τρόπο τον οποίο αντιμετώπιζε τους ε, πρόσφυγες, δεν θα είχαμε προβλήματα. Ε, έχουν περάσει αρκετά χρόνια τώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε τα μαθήματα ε, αυτών των περιπτώσεων και της περίπτωσης της Ουγγαρίας συγκεκριμένα. Το θέμα των προσφύγων, το θέμα των οικονομικών προσφύγων οπωσδήποτε είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το... και μια μεγάλη συζήτηση. Χαίρομαι πάντως που ξεκίνησε η συζήτηση. Χαίρομαι που άρχισε και πήρε το πρώτο βήμα, έκανε το πρώτο βήμα η Ευρώπη. Δεν θα σταματήσει εδώ η συζήτηση. Χαίρομαι πάντως που ξεκίνησε. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα ξανά τον λόγο στους επικεφαλείς των ομάδων με την αντίστροφη σειρά. Ο κύριος Μπορέλη ξεκινάει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία του εκφράζεσαι και του πληροφορήστε. Ε, αυτές είναι οι θεμέλοι, αυτά είναι τα θεμέλια επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και βεβαίω για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ των ουκάνευ προϋπόθεση είναι η μη χρήση της θανατικής ποινή. Εσείς μιλήσατε ε, για πραγματισμό κύριε Όρμπαν, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι έννοια έχει να μιλάτε ε, στους πολίτες ενός κράτους μέλους για θανατική ποινή εφόσον αυτή ρητά απαγορεύεται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρέπει να γίνονται βήματα προς τα πίσω αντί να κοιτάμε προς τα εμπρός ως ορθολογιστές και πραγματιστές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν θέματα και αξίες θεμελιώδη επί των οποίων ε, και με τα οποία κανείς δεν μπορεί ε, να παίξει για ε, ψηφοθυρικούς και εκλογικούς λόγους. Ευχαριστώ κύριε Μπορέλη. Κυρία Χάρμς. Είμαστε τελικά οι πολίτες της ε, Ουγγαρίας είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν αυτά που τους λέει ο κύριος Όρμπαν. Εγώ θεωρώ, γιατί ξέρω κάτι λίγα από την Ουγγρική ιστορία, πως οι Ούγγροι γνωρίζουν γιατί είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ελευθερίας και κατά αυτά τα οποία ε, μας παρουσιάσατε εσείς ε, και τον εθνικισμό αυτό. Πρέπει όμως να μας ανησυχεί όλους. Και εδώ θα συμπεριλάβω και τον κύριο Βέμπερ. Ότι στον, στο ερωτηματολόγιο αυτό συμβαίνει κάτι επικίνδυνο για την Ευρώπη. Γιατί δεν γίνεται ε, μόνο με μια γλώσσα προσβλητική αλλά με μια γλώσσα η οποία πραγματικά προκαλεί και συνδέεται με μεθόδους οι οποίες στη δική μου χώρα ε, χρησιμοποίησαν οι εθνικοσοσιαλιστές και έφεραν όλα αυτά τα κακά σε ολόκληρη την Ήπειρο. Και άρα θα πρέπει να είμαστε σε θέση στην Ευρώπη το 2015 από κοινού να κάνουμε κάτι. Αυτό ισχύει και για την Ουγγαρία και για άλλους ε, ε, που έχουν παρόμοια προβλήματα. Ευχαριστώ κυρία Τσίμερ. Κύριε Όρμπαν, θέλω να διαφωνήσω μαζί σας. Κανείς εδώ δεν ασκεί κριτική στην Ουγγαρία. Κανείς δεν ασκεί κριτική σε έναν λαό. Ασκούμε κριτική στη δική σας πολιτική, στις δική σας δηλώσεις, στο δικό σας άτομο, στο παιχνίδι που παίζετε για πολλωστή φορά. Έχουν εντύπωση πως έρχεστε εδώ πέρα γιατί θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να στείλετε το μήνυμα στο εσωτερικό ότι εγώ, ο Πρωθυπουργό, υπερασπίζομαι τη χώρα μας από αυτούς τους φοβερούς Ευρωπαίους βουλευτές ε, που ολοκριτική μου ασκούν. Σε, σε εσάς ασκούμε κριτική, όχι στους πολίτες της ε, χώρας σας. Θέλουμε να μπορούν να αποφασίζουν ε, οι πολίτες σας όπως και όλοι οι υπόλοιποι για το μέλλον τους. Θέλουμε να ε, υπάρχει η ίδια αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες όπως κάνουμε και εμείς. Αλλά δεν θέλουμε να υπάρχουν ερωτηματολόγια στα οποία ε, επικρατεί κινησμός. Αυτό το οποίο μας λέτε εδώ πέρα είναι σκέτος κινησμός. Δεν έχει ούτε μία σχέση με δημοκρατία και απορρίπτουμε αυτές τις θέσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Φερχόφστατ. Θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να προσέξει ιδιαιτέρως αυτά τα οποία λέει ο κύριος ε, ε, Όρμπαν ε, στην δευτερολογία του, στην απάντηση που έδωσε και ενδεχομένως να προχωρήσετε αυτή την ιδέα σχετικά με την δημοκρατική διακυβέρνηση γιατί νομίζω ότι δεν μπορούμε ΣΑΗ να συζητούμε για τα θέματα αυτά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάσουμε σε ε, κάποιο αποτέλεσμα, να καταλήξουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε επα, ε, επαορίστο τη συζήτηση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, ε, δεύτερο σημείο, Δυστυχώ, δεν απαντήσατε κύριε Όρμπανα στις διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν επί, των ε, ερωτήσεων. Ο κύριο Τίμερμαν, μάλιστα σα είχε αμφισβητήσει την ερώτηση 3, δεν απαντήσατε σε αυτό. Λέτε ωραία, τρομερό επιχείρημα, τεράστιο, δεν υπάρχουν φιλελεύθεροι πλέον στην ε, ε, Ουγγαρία. Ναι, υπάρχει το ΦΙΔΕΦ. ξέρετε τι είναι το ΦΙΔΕΦ ε, είναι η οργάνωση των φοιτητών, των φιλελευθέρων. Και ξαφνικά λέτε, άμα δεν υπάρχουν φιλελευθεροί, τι, χάσατε τις εκλογές και μετά γυρίσατε και θέλετε να γίνετε εθνικιστής έτσι ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε τις εκλογές. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Κέρκοπ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική και δύο είναι τα πιστεύα μου. Τα πιστεύω μου τα οποία ακόμα στηρίζω. Η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία για όσους ζουν σε χώρες όπου η Ουγγαρία να μπορούν να κάνουν να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις για το ποιος θα τους κυβερνά. Δεν άκουσα τίποτα εδώ απόψε που να μου κάνει να αλλάζω αυτή την πεποίθηση. Δεν μου αλλάζει. Δεν μου αρέσει η ρητορία των ε, αριστερών κυρίως εκπροσώπων και θα ήθελα να κλείσω απαντώντας στον κύριο Φερχόφστατ. Μας είπατε πως ήρθε η ώρα να κλείσει η συζήτηση για την Ουγγαρία. Θέλω να είμαι πολύ σαφής κύριε Φερχόφστα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Πίτελα. Ο κύριος Πιτέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Όρμπαν, μη λέτε ότι εμείς μιλήσαμε άσχημα για την Ουγγαρία και τους Ούγγρους, γιατί αυτό δεν ισχύει, είναι λάθος. Εμείς δεν θέλουμε να υποδείξουμε σε μια κυβέρνηση τι θα κάνει. Ούτε θέλουμε να επιβάλλουμε τίποτα σε οποιονδήποτε, εκτός από τον σεβασμό των θεμελιωδών ε, αρχών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν πάσχουμε από ορμπανίτιδα, δηλαδή ένα είδος αλλεργίας σε εσά. Δεν έχουμε τίποτα προσωπικό με εσά, απολύτως τίποτα. Θέλουμε να συζητήσουμε μονάχα ε, επί πολιτικής βάσεως ε, για την ε, μετανάστευση. Τα, τα των πολιτικών αγώνων δεν μας απασχολούν αυτή τη στιγμή εδώ. Αυτό που μας απασχολεί όμως είναι η θανατική ποινή. Είναι η ιδέα μιας μη ελεύθερης δημοκρατίας. Εσείς είστε ελεύθερος να, λέτε ό,τι θέλετε, αλλά πρέπει να πείτε όμως και στους πολίτες σας ότι με τον τρόπο αυτό ανοίγετε το, το δρόμο για μια εξέλιξη που θα οδηγήσει την Ουγγαρία εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρέπει να το πείτε αυτό. Οδηγείτε την Ουγγαρία εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κύριε Όρμπαν. Κύριε Βέμπερ, σας ευχαριστώ για την συζήτηση, για την ανταλλαγή των απόψεων. Πρέπει να πω πως οι αριστεροί σε πολλούς τομείς άσκησαν κριτική, όπως κάναμε και εμείς, αλλά υπάρχουν πράγματα που δεν ισχύουν. Δηλαδή η κυρία Χάρμς την έκανε με τις μεθόδους των Ναζί, η κυρία Τσίμερ μετά μας είπε πως ε, πρέπει να τελειώσει αυτή η συζήτηση. Μα εσείς ζητήσατε να γίνει συζήτηση περί Ουγγαρίας. Η δικιά σας ομάδα το ζήτησε. Κάποια στιγμή δηλαδή να σταματήσουν οι υπερβολές. Εν τω μεταξύ ακούσαμε λίγα πράγματα για το γεγονός το οποίο ανέφερε ο κύριος Όρμπαντ, πως η, ο κύριος, η Ουγγαρία είναι υποδειγματική χώρα στην υποδοχή προσφύγων. Πολλοί από αυτούς που μίλησαν δεν δέχονται πρόσφυγες. Και κύριε Όρμπαν πρέπει να πω κάτι στο θέμα των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα στην Ευρώπη. Επιτρέπεται. Αλλά η ελευθερία του λόγου συνδέεται πάντα με ευθύνη. Αυτά πάνε μαζί. Και όταν μιλάμε στην συζήτηση πρέπει να σκεφτούμε τι έχουμε κατακτήσει ως πολιτισμό σε αυτή την Ήπειρο, ότι το κράτος δηλαδή δεν μπορεί να σκοτώνει. Αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε και εδώ πέρα συμφωνούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί. Κύριε Τίμερμανς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποια σχόλια να κάνω για τα όσα ακούστηκαν. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον να ακούει κανείς πόσο έχει πετύχει σε οικονομική ε, κατάσταση στην Ουγγαρία και ξέρω πως ο κύριος Ορμπάν έχει πετύχει μερικές από τις πιο ε, εντυπωσιακέ εκλογικές ε, νίκες και αυτό είναι προς τιμή του. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως το κράτος δικαίου, όσο συντριπτική να είναι και η πλειοψηφία μιας κυβέρνησης, μπορεί να διακυριευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ως ε, πρόφαση την οικονομική άνθηση μιας χώρας για να ε, δηλώσει πως δεν χρειάζεται να σέβεται το κράτος δικαίου. Χαίρομαι που ακούω από ιστορίες οικονομικών επιτυχιών, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τη συζήτηση που γίνεται για το κράτος δικαίου. Η συζήτηση αυτή, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει να κάνει με πολιτικές κομματικές. Το καταλαβαίνω πως για εσάς ίσως αυτό είναι επιθυμητό, αλλά για εμάς δεν πρόκειται εδώ για συζήτηση κομματικού περιεχομένου. Ε, κάποιοι κατέταξαν στα αριστερά του φιλελευθέρου σήμερα, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μάλλον εκτός συζήτησης. Εν πάση περιπτώσει, είμαι σαφέστατα υπέρ της ελευθερίας του λόγου. Είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες, τις οποίες στηρίζουμε, είναι μία από τις αξίες ε, για τις οποίες όταν ήταν στην αντιπολίτευση ε, ο κύριος Όρμπαν έδωσε τεράστιες μάχες όσο ακόμα ε, καθεστώς ήταν ο κομμουνισμός τότε που ήταν φιλελεύθερος άλλωστε. Όμως η ελευθερία του λόγου περιορίζεται από το κράτος δικαίου. Εάν μου πεις πως θέλω να κάνω μια συζήτηση για την κατάργηση της θανατικής ποινής βεβαίως και μπορεί να το συζητήσεις αλλά πρόταση για την κατάρρευση θανατικής ποινής, με συγχωρείτε για την επαναφορά της ε, θανατικής ποινής, αποτελεί παραβίαση ε, διεθνών υποχρεώσεων. Ο Πρωθυπουργό και Ευρωπαϊκών Υποχρεώσεων πως είναι σύμβατο με την ε, ιδιότητα του μέλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Πρωθυπουργό κ. Όρμπαν είπε πως δεν έχει καμία πρόθεση να υποβάλει τέτοιου είδου πρόταση για την επαναφορά της Αντικής ποινής. Λοιπόν, αν δεν έχετε την πρόθεση να υποβάλλετε τέτοια πρόταση, γιατί γίνεται η συζήτηση. Υπάρχει κάποιος λόγος. Καμιά φορά και εγώ μπορώ να απευθύνω ρητορικέ ερωτήσεις. Δώστε μου αυτό το δικαίωμα. Τέλος, αν γίνει συζήτηση. Και σέβομαι κύριε Όρμπαν πως ήρθατε στην Ολομέλη γνωρίζοντας το τι θα ακούσετε. Ήρθατε εδώ να υπερασπιστείτε τη θέση σας και εγώ ως Δημοκράτη σέβομαι τη βούληση σας αυτή, αλλά θα σεβόμουν περισσότερο τη θέση σας αν οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα έπρεπε να παρουσιάζονται ως καρικατούρα έτσι όπως κάνατε εσείς σήμερα. Πού στις προτάσεις μας κύριε Πρωθυπουργέ λέμε πως χρειάζεται να ανοίξουμε τις πόρτες στους μετανάστες και στη μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποιο σημείο βρίσκεται. Θα ήθελα να μου το δείξετε. Πού στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετανάστευση που παρουσιάσαμε προτείνουμε ελευθερία για όλους τους οικονομικούς μετανάστες να έρθουν στις χώρες μας. Σε ποιο σημείο. Αντίθετα, εμείς αυτό που θέλουμε είναι μια πολύ πιο στεναρή πολιτική έτσι ώστε όσοι δεν έχουν δικαίωμα σε άσυλο να επιστρέφουν στις χώρες τους. Αυτό είναι κομμάτι αναπόσπαστο των προτάσεών μας. Αν μιλάμε για ποσοστώσεις, μιλάμε για ποσοστώσεις για πολύ περιορισμένες σοβαρές περιπτώσεις και υποθέσεις που απορρέουν από μια σοβαρή σύραξη. Γιατί οι περισσότερες αιτήσει ασύλου προέρχονται από ανθρώπους που φεύγουν από τη Συρία ή την Αιθιοπία όπου ξέρουμε τι συμβαίνει. Αλλά μιλάμε για ένα πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων και θα ήταν πολύ επιβοηθητικό για τη συζήτηση να μην προσφέρουμε καρικατούρες των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί καλό είναι να γνωρίζει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Κοινωνία ποιες είναι οι προθέσεις μας. Και κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους ανθρώπους μαζικά να καταφθάνουν στην Ευρώπη όταν δεν έχουν, δεν χρήζουν ασύλου. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να μείνουν στις χώρες τους. Να τους βοηθήσουμε να μείνουν στις περιοχές στις οποίες ανήκουν. Και όλα αυτά αποτελούν κομμάτια της προτάσης, των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το λέω με τέτοια ένταση, γιατί πιστεύω ότι η συζήτηση για τη μετανάστευση θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και σαφεί για το ποιε είναι οι προθέσει μα και ποια είναι τα σχέδιά μα. Όλοι. Η έκκληση που απευθύνω από το βάθη τη καρδιά μου στην ε, Ουγγρική κυβέρνηση και σε όλου είναι σα παρακαλώ πολύ, τα σχέδια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μην τα βλέπετε ω καρικατούρε, γιατί εμεί, αυτή τη στιγμή για την πάταξη τη λαθρομετανάστευση, είμαστε στο ίδιο, στην ίδια πλευρά του μετόπου. Όμως, θα πρέπει να είμαστε σε πλήρη συμμόρφωση με τις κοινέ μας αξίες. Αξίες τις οποίες όταν είστε νέος ε, υπερασπιστήκατε και εσείς κύριε Πρωθυπουργέ όταν είχατε απέναντι σας κομμουνιστές. Είναι οι αξίες που είναι κοινέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπαίνετε στη συζήτηση γιατί ξέρετε σαφέστατα πως έχουμε το δικαίωμα να συζητάμε μεταξύ μας τις αξίες αυτές. Δεν μπορείτε να πείτε ότι κανείς μπορεί, από άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συζητήσει τι γίνεται στη χώρα μου. Όχι. Ίσα ίσα. Αυτό ακριβώς σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είμαστε μέλη. Θα πρέπει να συζητάμε τα θέματα αμφότερων με σεβασμό, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιον από τη συζήτηση ε, από κάποιο άλλο κράτος μέλος επειδή δεν είναι υπήκο του κράτους αυτού. Ανήκουμε σε μια κοινότητα αξιών. Και θα ήθελα να κλείσω συζητώντας για τις πολύ δύσκολες περιπτώσεις των ε, προσφύγων. Εγώ γνωρίζω καλύτερα, καλύτερα την κατάσταση στην Ολλανδία και ξέρετε πόσα ονόματα πια θεωρούνται Ολλανδικά. Ε, σας, τότ, για παράδειγμα, είναι πολύ πετυχημένα οι Ολλανδοί στην Ολλανδική κοινωνία και είναι παιδιά ανθρώπων που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν ε, την Ουγγαρία όταν η Σοβιετική Ένωση ε, το 1956 κατέπνιξε την ανάγκη για ελευθερία των Ούγγρων και εγώ χαίρομαι που τον Τότ, τον Σάτς και τον Νίμιτς τον έχω στη χώρα μου και θεωρώ πως είναι κομμάτι της Ολλανδικής κοινωνίας και της κοινωνίας μας κοινωνίας αξιών και κατάφεραν να έρθουν στη χώρα μας για το 1956 οι Ευρωπαίοι ήξεραν πως οι απελπισμένοι που εγκαταλείπουν την Ουγγαρία χρειάζονται καταφύγιο. Άνοιξαν τα σπίτια τους, τις καρδιές τους, τις κοινωνίες τους και αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι ένα παράδειγμα που αποδεικνύει το τι ακριβώς σημαίνουν οι ευρωπαϊκές αξίες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Συμβούλιο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε Σόλτσο. Κύριε Πρόεδρε Τίμερμαντς, κυρίες και κύριοι Βουλευτέ, πραγματικά ελπίζω ότι αυτή η σημερινή πρόσωπο με πρόσωπο ανταλλαγή ε, απόψεων ε, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ο ένας καλύτερα τις ε, θέσεις του άλλου. Άκουσα με πολύ προσοχή όλο το φάσμα των απόψεων που εξεφράστηκαν στη διάρκεια της συζητήσεως. Όπως ε, είπα και στην ε, αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία ένωση ε, ε, θεμελιωδών ε, αξιών, τις οποίες μοιράζονται όλοι και που ισορροπούν και αποτελούν βάση των θεσμικών οργάνων και της θεσμικής τοποθέτησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προϋπόθεση ή μία από τις προϋποθέσεις είναι η μη ύπαρξη θανατικής ποινής. θενατικης αξίες. Δεν είναι δυνατόν βεβαίως να απαγορεύσουμε μια συζήτηση, οποιαδήποτε συζήτηση συζήτηση. Ταυτόχρονα όμως ευελπιστούμε ότι η έκβαση αυτής της συζήτησης θα επιβεβαιώσει ξανά τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία της έκφρασης επίσης είναι ε, βασική αρχή, αλλά έχει και κάποια όρια. Ας πούμε, απαγορεύονται ο ε, εξτρεμιστικός, ακραίος λόγος. Είχαμε σήμερα μία συζήτηση ε, και Όλοι είπαν ότι η αρχή, το δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές, ελεύθερες δυνατότητα εξέβρεση εργασίας και τα λοιπά είναι βασικές ε, ε, αξίες. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, όταν παίρνει κανείς μέτρα έτσι ώστε να προστατέψει τις δικές του αξίες γιατί κάποια μέτρα είναι υπερβολικά ακραία. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μέχρι να πείσουμε ένα τον άλλον. Έστω και αν αυτό δεν συμβεί σήμερα. Κυρίες και κύριοι, όπως ε, ήδη έχω αναφέρει, μιλάω εδώ ως Προεδρεύουσα ε, του Συμβουλίου και επομένως εξ ε, και των 28 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια δύσκολη δουλειά και μάλιστα μια και το θέμα που συζητήθηκε σήμερα εδώ δεν έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο, άρα δεν έχω μεγάλη ε, ε, ε, γκάμα επιλογών. Ωστόσο δεσμεύομαι να μεταφέρω τη συζήτηση αυτή στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι, τελείωσε η συζήτηση.